Καλημέρα σας, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καθίστε παρακαλώ. Για να αρχίσει ε, το δεύτερο μισό της σημερινής μας συνεδρίασης, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. I open the... Ευχαριστώ πολύ. Άρχεται λοιπόν η απογευματινή συνεδρίασή μας της 24 Ιανουαρίου. Βασικό σημερινό θέμα για το απόγευμα είναι ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Τόμισλαβ Ντόντσεφ, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης αρμόδιο για τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την οικονομική πολιτική. είναι και Προεδρεύων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μας μιλήσει για τις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η χαρά μου Βουλγάρα να υποδέχομαι τον Αντιπρόεδρο της Βουλγαρικής Κυβέρνησης στην Επιτροπή μας για να μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας για την πολιτική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη. Καλώς ορίσατε κύριε Ντόντσεφ, με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω εδώ. πώς ε, θα έχει η διαδικασία ως ήθιστε. Θα ακούσουμε τον κύριο Ντόντσεφ ε, που θα μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Προεδρίας. Στη συνέχεια θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε ερωτήσεις για να ανταλλάξουμε απόψεις αρχής γενομένης από ε, τις ερωτήσεις των συντονιστών των πολιτικών ομάδων. Ωραία. Χωρίς περιττέρω καθυστέρηση, κύριε Ντόντσεφ, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα προσπαθήσω να μιλήσω βουλγαρικά. Όχι μόνο γιατί είναι καλύτερα τα βουλγαρικά μου σε σύγκριση με τα αγγλικά μου, αλλά και για να σας δώσω την ευκαιρία να ακούσετε την όμορφη μελωδία της βουλγαρικής γλώσσας. Επίσης, πρέπει να δείξουμε ότι μπορούμε να μεταφράσουμε την ε, περιφερειακή πολιτική και την πολιτική συνοχή σε όλες τις πιθανές γλώσσες. Και παρακαλώ, προετοιμάστε τα ακουστικά σας. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο σκοπός της σημερινής ε, ακρόσης είναι να παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Βουλγαρικής ε, Προεδρίας και πιο συγκεκριμένα αυτές που σχετίζονται με τη συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Ωστόσο, θα ήθελα να μη σταθώ στο πρωτόκολλο Επιπροσθέτω της ε, σύντομης παρουσίασής μου, θα ήθελα να έχουμε μια ειλικρινή συζήτηση, όχι μόνο επί των προτεραιοτήτων μας ως Προεδρία, κυρίως στον τομέα της πολιτικής συνοχής, αλλά και για το μέλλον του κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος. Γιατί πιστεύω ότι μόνο όσοι γνωρίζουν που πάνε έχουν μέλλον. Ορίστε λοιπόν οι τέσσερις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας, το μέλλον της Ευρώπης ε, και των νέων, οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, οι ευρωπαϊκές προοπτικές ε, και η συνδεσιμότητα των Δυτικών Βαλκανίων, ασφάλεια και σταθερότητα σε μια ενωμένη και ισχυρή Ευρώπη και τέταρτον ψηφιακή οικονομία και οι δεξιότητες που χρειάζονται για το μέλλον. Αυτές οι προτεραιότητες αντικατοπτρίζουν ε, τις ε, προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζουμε. Δεν θέλω να υποτιμήσω τις άλλες προτεραιότητες όσο σχετίζονται με το μέλλον των νέων, με την ψηφιακή οικονομία. Αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι η συγκεκριμένη προτεραιότητα που έχει να κάνει με την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Πριν 20 χρόνια είχαμε πόλεμο στα Βαλκάνια και οι πληγές ε, του πολέμου δεν έχουν απολωθεί ακόμη. Όλοι μας ε, τότε και η Βουλγαρία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στέκονταν και παρακολουθούσαν χωρίς να μπορούν να κάνουν τίποτα. Ένα νέο τέτοιο σενάριο μπορεί να αποφευχθεί μόνο αν δώσουμε ξεκάθαρη πολιτική προοπτική στους γειτονές μας στα Δυτικά Βαλκάνια. Γιατί εκεί όπου υπάρχει ευημερία και κοινέ αξίες μας έχει διδάξει η ιστορία ότι δεν προκύπτουν πόλεμοι. Λόγω της ε, ιδιαιτερότητας ε, αυτής της ε, περιοχής η Βουλγαρία θέλει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Θέλω να ξεκινήσω την παρουσίασή μου με την πολιτική συνοχής λέγοντας ε, ότι ενδομονώ για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ξέρω ότι ως ένα βαθμό αυτό είναι κλισέ, όμως περιλαμβάνει πολύ καλά την ε, περίοδο της Βουλγαρικής Προεδρίας ε, στο πνεύμα της κινέζικης της αρχές κινέζικης κατάρας μακάρι να ζει σε ενδιαφέροντες καιρούς. Αντιμετωπίζουμε τις παραδοσιακές προκλήσεις, που γνωρίζουμε πολύ καλά. Σχετίζονται και με την ανάγκη να φέρουμε πιο κοντά τις χώρες, αλλά έχουμε και νέες προτεραιότητες, σχετικά νέες, που έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Από την άλλη πλευρά, η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση προϋποθέτει πολιτικές ε, και οικονομικές προκλήσεις. Είναι σημαντικό να τονίσουμε τον τεράστιο κίνδυνο το κίνδυνο του να χάσουμε την αίσθηση ότι έχουμε ένα κοινό στόχο. Να σας υπενθυμίσω, πριν 10 χρόνια η στόχοι μας ε, ήταν να ξεπεράσουμε τους παγκοσμίους ανταγωνιστές μας. Να είμαστε καλύτεροι στην καινοτομία και στην έρευνα. Είχαμε αυτοπεποίθηση να ανταγωνιστούμε με τις άλλες χώρες. Τώρα, με πάση ειλικρίνεια, πρέπει να παραδεχτούμε ότι ενίοτε ε, μοιάζει, μοιάζουν οι δράσεις μας ε, σαν ε, δράσεις διαχείρισης κρίσεων και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και μια νέα κρίση. Δεν θα ήθελα όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ένα επιτελείο διαχείρισης κρίσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδειχθεί ικανή να πράξει κάτι τέτοιο. Όμως, πέρα από την κρίση, θα πρέπει να θετούμε και εμείς υψηλότερους στόχους και επιστρέφω στην πολιτική συνοχή. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι σύμφωνα με πολλούς εμπειρογνώμονες αυτή είναι η πιο επιτυχή και η πιο μεταρρυθμισμένη και σχολιασμένη ευρωπαϊκή πολιτική. Ταυτόχρονα η υιοθέτηση της πολιτικής αυτής από τους πολίτες μας ε, ε, δεν γίνεται αυτόματα. Φυσικά θα έχουμε και τη συζήτηση για το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και την πολιτική συνοχής που αναλογεί στο 1 τρίτο του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Θα πρέπει ε, να απαντήσουμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση. Εδώ κατά νου τη μετανάστευση και την ασφάλεια θα πρέπει να προωθήσουμε και τη σύγκληση μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ισχυρή μόνο αν όλοι οι πολίτε από το Ελσίνη και μέχρι την Αθήνα και από τη Λισαβόνα μέχρι το Βάρνα έχουν το ίδιο επίπεδο ζωή, το ίδιο επίπεδο διαβίωση. Βέβαια, είναι μακρινό αυτό ο στόχο γιατί ε, παρά τι επενδύσει που έχουν γίνει, οι πιο φτωχοί εξακολουθούν να είναι 10 φορέ φτωχότεροι από του πλουσιότερου. Αυτό σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς, σύμφωνα με άλλους υπολογισμούς, μπορεί το χάσμα να είναι και 20 φορές μεγαλύτερο. Η πολιτική συνοχή λοιπόν χρειάζεται να εξισορροπήσει κάποιες ανισορροπίες της ε, ενιαίας αγοράς, όμως ταυτόχρονα μαζί με τη σύγκληση θα πρέπει να καταστήσει και πιο ισχυρή, πιο ανταγωνιστική την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλύτερη για τους πολίτες. Και εδώ έρχεται η πρώτη μου ανησυχία. Σχετίζεται με την απουσία μια ευρύτερη συζήτηση για τι κοινέ μελλοντικέ μα προοπτικέ. Πρόκειται να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για το μελλοντικό πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο χωρί παράλληλη συζήτηση για την Ευρώπη του 2030. Ποιε είναι οι κοινέ μας προτεραιότητες. Πώς θα πετύχουμε βιώσιμη σύγκληση. Πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταστεί παγκοσμίω παίκτη. Ή αν προσπαθήσουμε να φέρουμε τη συζήτηση σε πιο τεχνικό επίπεδο, ποιες θα είναι οι νέες θεματικές ε, και οι αρχές της θεματικής συγκέντρωσης στους μελλοντικού κανονισμούς που θα αφορούν τα Ευρωπαϊκά Διορθωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε μόνο αν ξέρουμε προς τα που κατευθυνόμαστε. Βάσει της εμπειρίας μου δεν είναι ορθή πρακτική να σχολίζουμε την προπολογισμό και την κατανομή του προπολογισμού αν δεν ξέρουμε τους στόχους μας, τις προτεραιότητες και τις πολιτικές μας. Και εδώ αξιότιμα μέλη προτείνω και απευθύνω έκκληση σε εσάς πριν κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για την αποτελεσματικότητα του προπολογισμού των εργαλείων των προγραμμάτων και των αριθμών να μιλήσουμε για στόχους και προτεραιότητες. Ας είμαστε επιμελεί και α κάνουμε τους λογαριασμούς μας. Όμως, ας μην ξεχνάμε να έχουμε και οράματα, να μην είμαστε απλοί λογιστές. Η δεύτερη ανησυχία μου βασίζεται στο γεγονός ότι για πολλούς λόγους και κυρίως ε, λόγω Brexit θα πρέπει να μάθουμε πώς θα πετύχουμε περισσότερα με λιγότερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα Δεν μπορεί να το μαγικό ραβδί, γιατί ε, δεν ε, ασκούμε την αλχημία. Πρέπει να, προβλε... μετατρέψουμε αυτή τη φόρμουλα σε συγκεκριμένο μηχανισμό, μεθοδολογία ή προσέγγιση. Υπάρχουν διάφορα βασικά σημεία. Καταρχήν θα πρέπει να επενδύσουμε σε τομείς με υψηλή προσθεμένη αξία. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Παρ' όλα αυτά, το σημείο αφετηρίας μας θα πρέπει να είναι η κοινή κατανόηση για το τι εννοούμε με το υψηλή προστιθέμενη αξία. Το δεύτερο σημείο είναι ότι πέρα από τις επενδύσεις σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας θα πρέπει να εξετάσουμε και επενδύσεις σε μεταρρυθμισμένους τομείς και να εγγυηθούμε την αποδοτικότητα κάθε επένδυσης. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα και να υπάρξουν και μεταρρυθμίσεις. Βέβαια, αν θέλουμε να πετύχουμε περισσότερα με λιγότερα, θα πρέπει να βελτιστοποιήσουμε τη ροή των επενδύσεων. Κάτι που αναπόφευκτα σχετίζεται με την ε, ριζική απλούστευση των κανόνων. Στα τέλη του περασμένου χρόνου, σε εθνικό επίπεδο, αναλύσαμε το επίπεδο των ε, ελέγχων ε, που υλοποίησαν οι διαχειριστικές αρχές. Τα αποτελέσματα ήταν ε, ιδιαίτερα ενισχυτικά. Διαδικασίες ε, που αφορούσαν 70 ελέγχους απαιτούσαν πάνω από 46 συνοδευτικά έγγραφα από τους δικαιούχους. Και αυτή είναι η γενική εικόνα, δεν είναι εθνική ιδιαιτερότητα. Μάλιστα, Αυτά συνέβησαν παρά τι συστηματικέ προσπαθίε μας να, ζητάμε πράγματα, να μην ζητάμε πράγματα που δεν χρειαζόμαστε. Αυτό δεν οφείλεται σε έλλειψη διοικητική ικανότητα. Έχουμε επενδύσει πολλά στου ανθρώπου αυτού και έχουν αποδείξει την εμπειρία τους. Όμως το θέμα είναι Μήπω ε, κάποια στιγμή οι ελεγκτέ μας πούν ότι χρειάζεται κάποια δημοσιονομική διόρθωση κάποια μέρα ή μήπω ε, θα παραλείψουμε κάποιο έγγραφο και αν ε, γίνει κάποιο λάθος ποιο θα φταίει. Αυτό δημιουργεί δυσκολίε και για του δικαιούχου αλλά και για τις αρμόδιες αρχές. Πιστεύω λοιπόν ότι χρειαζόμαστε Κάποιε επαναστατικέ λύσει. Εγώ προέρχομαι από την Ανατολική Ευρώπη, όπου είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αν χρειαζόμαστε μια επανάσταση, θα έχει να κάνει με την απλούστευση των κανόνων. Μπορούμε να πετύχουμε την πραγματική απλούστευση μόνο αν είμαστε θαραλέοι και αν αλλάξουμε την προσέγγιση μας. Αντί να επικεντρωνόμαστε στα έγγραφα, να επικεντρωθούμε στα αποτελέσματα και στους στόχους. Πρέπει να απτύξουμε ένα νέο κουτί εργαλείων, ένα νέο toolbox ε, που θα έχει να κάνει με τον έλεγχο των εγγράφων. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ένα καλό έλεγχο. Πολλές φορές ε, μιλάμε και για ένα πολύ αυστηρό έλεγχο, αλλά εγώ νομίζω ότι ο έλεγχος θα πρέπει να είναι καταρχήν ευφυή. δεν είμαι σίγουρο ότι είναι η φιλοσοφική λήθο ε, τη μυστική τάξη το να κάνουμε περισσότερα με λιγότερα, αλλά τουλάχιστον μπορεί να είναι καταλήτη. Η Βουλγαρική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπίπτει με τις τελικές προετοιμασίες της νομοθετικής πρότασης της Κομισιόν για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε λοιπόν την πρόκληση της επίτευξης συνένεσης σε θέματα όπως ε, η εθνικοί συντελεστές χρηματοδότησης για την πολιτική συνοχή, σε προτεραιότητες και θεματική συγκέντρωση στην ε, πολιτική συνοχή, κριτήρια για ε, τις ε, εθνικές και κατανομές των κονδυλίων. Θα υπάρχουν έντονες συζητήσεις για αυτά τα θέματα, αλλά εδώ πρέπει να αναρωτηθούμε ως αφετηρία τι είδους πολιτικής θέλουμε μετά το 2020. Θα πρέπει να είναι μια πολιτική που να προωθεί τη σύγκληση και να ενθαρρύνει την ανταλλαγή κοινών αξιών ή θα είναι μια πολιτική που θα επικεντρώνεται σε κάποιες περιφέρειες ή θα πρέπει να καλύψει όλες τις περιφέρειες. Μήπως εμείς ως κράτη-μέλη θα έπρεπε να συνεισφέρουμε περισσότερο. Αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο αναμένω έντονες συζητήσεις και μήπως ε, κάτι τέτοιο ε, δεν θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη υπερθεροποίηση των φτωχότερων περιοχών που δεν θα μπορούσαν να σεβαστούν τις απαιτήσεις της χρηματοδότησης. Εγώ πιστεύω ότι αυτές ε, οι ερωτήσεις, αυτά τα θέματα θα καθορίσουν τη μελλοντική συζήτηση και θα είναι οι κύριες προκλήσεις για την Βουλγαρία στο πλαίσιο της Προεδρίας μας. Αυτά θα είναι τα θέματα που σκοπεύουμε να θέσουμε προς συζήτηση για την πολιτική συνοχή στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που θα λάβει χώρα στις 12 Απριλίου και στην ε, διάσκεψη στη Σόφια στις 8 Ιουνίου. Επιτρέψτε μου να εκφράσω την ελπίδα μου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι ένα ζωτικός εταίρος ε, στο να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις. Και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, η Βουλγαρία είναι μια ε, χώρα που τις βάζουν διάφορες ετικέτες. Είναι μια χώρα που έχει πετύχει πολλά τα τελευταία δέκα χρόνια μετά την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό οφείλεται όχι μόνο στην καλή βούληση και στη φιλοδοξία της, αλλά οφείλεται ιδίως στην εμπειρία που έχουμε κερδίσει από τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων και αναφέρομαι στις πρακτικές πτυχές. Επομένως, είμαι πεπισμένος ότι όλες αυτές οι ικανότητες, βάσει και των διδαγμάτων που έχουμε αντλήσει, από τη θέση ενός διαμεσολαβητή ειλικρινούς που επιζητά συμβιβασμό στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, μπορούμε να συνεισφέρουμε Ταυτόχρονα, φιλοδοξία μου είναι πως ε, όταν ε, χρειάζεται μπορούμε να είμαστε ηγέτες ή μπορούμε να παράγουμε νέες ιδέες. Γιατί χρειαζόμαστε νέες ιδέες. Νέες ιδέες, φρέσκες ιδέες τις αποκαλούμε στη Βουλγαρία που οδηγούν σε ένα κοινό μας μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, στα βουλγαρικά και στα αγγλικά. Η Πρόεδρος ε, μας εμπνέει η ομιλία σας. Θα δώσω αμέσω το λόγο στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων, αρχής από τον κύριο Φανίστερ Ρόι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πολύ Υπουργέ που ξανάρθατε ε, εδώ στην Επιτροπή μας, όπου η συνοχή, η συνεκτικότητα και η ελεγγύη στην Ευρώπη είναι πρωταγωνιστικά. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σας. Βεβαίως η Προεδρία του Συμβουλίου πολλά συντονίζει, άλλα διοργανώνει και σημαντικά για τα όσα μας αφορούν εμάς και αφορούν και τη χώρα σας. Εξού και πολιτική συνοχής. Δεν χωρά καμία αμφιβολία ότι είναι προτεραιότητα για σας. Και χαίρομαι που μετά την Μαλτεζική ε, Προεδρία ε, είναι καλό που συνεννοήθηκαν οι υπουργοί μετά από μια υπουργική απόφαση ε, να επιληφθεί ε, το Συμβούλιο Υπουργών Γενικών Υποθέσεων. Και στο Κοινοβούλιο είχαμε την έκθεση Westphal για το μέλλον της πολιτικής συνοχής και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων ευθυγραμμίζονται πάρα πολύ με τα όσα εμείς εδώ συζητούμε. Άρα πριν το επόμενο Συμβούλιο Γενικών Υπηθώσεων, δεν, γιατί δεν υπάρχει Συμβούλιο Υπουργών Συνοχής αυτό καθ' αυτό, ασχολείται το Συμβούλιο ε, Γενικών Υποθέσεων. Ε, ελπίζω να θέσετε αυτό το θέμα της συνεκτικής πολιτικής και στην πολιτική συνοχής. Ωραίες οι προτεραιότητές σας. Έχω μερικά σημεία να σχολιάσω σε σχέση με τα όσα είπατε. Πρώτον, Αναφερθήκατε ε, σε μια επανάσταση. Δύο φορές ε, χρησιμοποίησατε τη λέξη επανάσταση και δεν μπορεί να έχω κάνει λάθο αφού την επαναλάβατε. Επανάσταση κυρίως στον τρόπο με τον οποίο δρούμε και διαχειριζόμαστε ε, τα πράγματα και δίνουμε αρμοδιότητες και ευθύνε που θα πρέπει και, και λογοδοσία για να βρούμε την ισορροπία που χρειάζεται. Προτάσεις κάνετε, γιατί κάνετε ερωτήσεις και οι ερωτήσεις ζητούν απαντήσεις. Η Προεδρία τι θα κάνει για να τα υλοποιήσει όλα αυτά και να γίνουν πραγματικότητα. Εγώ ιδέες έχω πολλές. Για την επόμενη φάση μετά το 2020 μπορεί να έχουμε και λιγότερα χρήματα για τη συνοχή. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για τη συγχρηματοδότηση και ποιος θα ελέγχει Τώρα ελέγχουν τα κράτη-μέλη, ελέγχει και η Ευρώπη. Υπάρχει ένας κύκλος. Υπάρχει κάτι που μπορεί να ακούγεται εδώ επαναστατικό, αλλά τι προτείνετε. Ε, ε, κινούμαστε προς την κατεύθυνση ε, του κανονισμού Omnibus, το αναφέρατε κι εσείς, για την απλούστευση, αλλά μπορεί να χρειαστούν και μεγαλύτερα βήματα. Ενδιαφέρομαι λοιπόν, τι είναι αυτή η επανάσταση, τι προτάσεις θα φέρετε συγκεκριμένα. Πρώτη ερώτηση. Ερώτηση δεύτερη για τον κοινωνικό πυλώνα, λέτε εδώ στο έγγραφό σας ότι θα προωθήσετε ε, την υπόθεση αυτή και θα κάνετε προτάσεις για την κοινωνική Ευρώπη και για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, λέτε. Μα εκεί ακριβώς η Επιτροπή Συνοχής, η δική μας Περιφερειακή Επιτροπή, παρακολουθεί τις εξελίξεις. Το Κοινωνικό Ταμείο στην Ευρώπη έχει πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό από τα ε, χρήματα της συνοχής από ότι ποτέ στο παρελθόν. Είχαμε 20-23 και τώρα είμαστε στο 27%. Και θέλω να απευθύνω μια έκκληση το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που χρηματοδοτεί σχολεία, έργα υποδομής, ε, σπίτια και κοινωνικά και άλλα θα πρέπει να είναι ενωμένο με το Κοινωνικό Ταμείο, να μην το διαχωρίσουμε γιατί κάποιοι θέλουν να το παραγωνίσουν τελείως το Κοινωνικό Ταμείο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Να μην χάσουμε αυτή τη συνέργεια, αυτή την υπεραξία, ε, την τρομερή που έχουμε τώρα στην περιφερειακή πολιτική με τα δύο ταμεία θα πρέπει να παραμείνει αυτό στις πόλεις, περιφέρειες και στις χώρες. Ρωτάτε αν διαχειριζόμαστε την κρίση. Όχι. Καμιά φορά καλείστε να διαχειρίζετε και κρίσεις. Αλλά το βασικότερο είναι να διατηρήσετε κάποια πράγματα που πηγαίνουν καλά. Και πολλά πράγματα στο σχεδιασμό της περιφερικής πολιτικής λειτουργούν καλά. Να μην πεταχθεί στην άκρη ε, το ταμείο αυτό το κοινωνικό. Και τέλος, μιλάτε για την προβολή, για την δημοσιότητα. Αν δείτε τις δημοσκοπήσεις, οι πολίτες καταλαβαίνουν τι κάνουμε, βλέπουν περισσότερα τι κάνουμε. Και στα εξωτερικά μας σύνορα, με την οικονομική ανάπτυξη και ανάκαμψη. ίσως θα πρέπει να παρουσιάζουμε καλύτερα τα αποτελέσματά μας και στην ε, χώρα σας και στις ελληνικές μας χώρες και εκεί θα πρέπει να αφήνουμε τα στέρια να λάμουν, δηλαδή τα στέρια της Ευρωπαϊκής Σημαίας. Να το προβάλλουμε, να δείχνουμε ότι είναι μια κοινή προσπάθεια και κοινό το αποτέλεσμα. Και αυτό δεν σημαίνει πολύ ε, συχνά. Ε, όλα τα κακά τα φορτώνουμε στην Ευρώπη και τα καλά δεν είμαι σίγουρος ότι τα πιστώνουμε στην Ευρώπη εμείς από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουμε τον Ιούνιο μια έκθεση στο Κοινοβούλιο όπου θα παρουσιάζουμε ε, αυτά τα καλά παραδείγματα και τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τελευταίο σχόλιο. Μας καλέσετε για τη συνεδρίαση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εμεί δεν μπορούμε να πάμε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, αλλά τον Ιούνιο θα γίνει μια σημαντική συνάντηση και περιμένουμε να μα προσκαλέσετε. Μια ευρύτερη αντιπροσωπεία τη Επιτροπής μα να συμμετέχουν εκεί σε αυτή τη διάσκεψη. Τη σημειώνουμε την πρόσκληση, γιατί είναι στι παραμονέ ε, της παρουσίασης των κανονισμών μάλλον και μετά την παρουσίαση των προτάσεων για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Συγχαρητήρια. Μα ε, μας χαροποιούν πάρα πολύ τόσα μας είπατε ως προτεραιότητες. Ευχαριστώ. Σοσιαλιστές και δημοκράτες. Η κυρία Βέστφαλ. <laughs> Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έπεσε σε μένα ο κλήρος τώρα να μιλήσω εξ ονόματος των σοσιαλιστών. Ας αρχίσω με το εξής. Μας καλέσατε κύριε Υπουργέ να είμαστε στο πλευρό σας παραστάτες στον αγώνα για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Μπορώ να σας πω απερίφραστα και ειλικρινά ότι κατά πλειοψηφία το Κοινοβούλιο πέρυσι αποφάσισε να βάλει τα θεμέλια σε μια έκθεση πρωτοβουλίας για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Και θα ήθελα να το πω αυτό ξεκάθαρα διότι στην παρουσίασή σας αναφερθήκατε ήδη σε κάποια από τα σημεία που μας απασχολούν και εμά. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή ξέρουμε και ποιε συζητήσει γίνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. θα πρέπει στο μέλλον όλες οι περιφέρειες να συμμετέχουν στην πολιτική συνοχή γιατί μας τα μπερδεύει λίγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό έχει να κάνει και με την αλληλεγγύη φυσικά. Και η αλληλεγγύη δεν είναι μόνο να δίνεις, αλλά να μπορείς και να παίρνεις. Και αν οι πλούσιες περιφέρειες δείξουν περισσότερη προθυμία να δώσουν περισσότερα χρήματα, αυτό είναι ευπρόσδεκτο. Αλλά αυτό σημαίνει αντίστροφα ότι υπάρχει και ανάγκη στις δικές μας περιφέρειες να ε, προωθούνται και αυτές και να ισχύονται. Λοιπόν, εμείς ως Επιτροπή και ως Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσαμε μεν ε, κατά πλειοψηφία τη διατήρηση της πολιτικής συνοχής και μάλιστα προς όλες τις περιφέρειες να είναι επιλέξιμες όλες. Βέβαια γνωρίζουμε ότι μετά το Brexit που μας λυπεί πάρα πολύ θα αλλάξουν τα πράγματα και θα χάσουμε ετησίως 12 με 13 δισεκατομμύρια από τον κουρβανά μας ενώ τα καθήκοντα και υποχρεώσεις δεν μειώνονται. Για να μην πω ότι αυξάνονται μάλιστα. Και πιθανόν να υπάρξει μείωση των πόρων αλλά με μέτρο γιατί και η πολιτική συνοχής έχει πολλές υποχρεώσεις. Μόλις επέστρεψα από μια διάσκεψη για την αστική πολιτική και πριν από δύο χρόνια ήμουνα και στη Σόφια για αυτό το θέμα. Παραμένει επιτακτική ανάγκη να ασχοληθούμε με τις πόλεις, γιατί ακριβώς στα αστικά κέντρα ε, ζουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ε, είναι πολλά τα κονδύλια που χρειάζονται και ανεξαρτήτως μεγέθους πόλης. Μιλήσατε και για την απλούστευση. Βεβαίω το γνωρίζουμε ότι οι διαδικασίε είναι πάρα πολύ περίπλοκε, όχι όμω σε όλε τι χώρε. Υπάρχουν και μερικέ χώρε όπου τα πράγματα γίνονται <clears throat> με ένα κλικ ε, στο ποντίκι του υπολογιστή. Ε, σε κάποιε άλλε χώρε είναι πολύ περίπλοκε οι διαδικασίε από την ε, υποβολή της αίτησης μέχρι τη χρηματοδότηση. Εκεί αποφασίσαμε ενδεχομένως να ακολουθήσουμε ένα καινούριο δρόμο ως κοινοβούλιο και να πούμε ότι στι περιφέρειες που πηγαίνουν καλά τα πράγματα δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να τα ανατρέψουμε αυτά. Ας αφήσουμε αυτά που λειτουργούν σωστά. Επίσης έχουμε την άποψη ότι σε κάποιους τομείς χρειάζεται μεγαλύτερη ευελιξία. Τι σημαίνει αυτό. υπάρχουν και απρόοπτα. Μπορεί μια περιφέρεια να λειτουργεί καλά και να υποστεί μια θεομηνία για να συγκλονιστεί ή να υπάρξει μια οικονομική καταστροφή. Να μπορούν να παρακρατούν ένα ποσό ε, τα μία συνοχής ε, για έκτακτες ανάγκες για να μπορούν επιγόντως να αντιδρούν. Επίσης, ε, νομίζω ότι είναι πλέον απαρχαιωμένο το σύστημα που είχαμε στο παρελθόν, όπου δίναμε γενικά χρήματα ε, σε όλους, όπως ένα ποτιστήρι που ποτίζει ε, παντού το ίδιο. Χρειάζεται μεγαλύτερη συγκέντρωση. Αλλά όλα αυτά είναι λεπτομέρειες. Το ουσιαστικό είναι να υπάρξει καν πολιτική συνοχή και να συνεχιστεί. Την περασμένη εβδομάδα συζήτησα με τον Επίτροπο Έτιγκερ. Ξέρω ότι είναι στο πλευρό μας, αλλά ακούγονται και άλλες φωνές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επικριτικές. Και για μας η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πολιτική συνοχή είναι ε, πραγματικά το... Ε, τσιμέντο που ενώνει ε, τα τούβλα στο οικοδόμημα. Η συγκολητική εκείνη η ουσία που μας κρατάει μαζί. Και χαίρομαι που είναι πολύ φίλοι της συνοχής και εσείς ως Προεδρία. Για να παραμείνει η πολιτική συνοχής κάτι που θα υπάρχει και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από την ECR, η κυρία Τόμασίτς. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ εκ μέρους της ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών θέλω να σας συγχαρώ για τη Βουλγαρική Προεδρία και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία το προσεχές εξάμεινο για την επίτευξη των προτεραιοτήτων σας. Χαιρετίζω ιδιαίτερα στην προτεραιότητα που αναφέρεται για το μέλλον της Ευρώπης και των νέων. Οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή. Τους επόμενους μήνες θα πρέπει να εργαστούμε στενά ε, έχουμε σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Ε, ξέρουμε ότι ε, οι περιορισμοί είναι αρκετοί ιδίω με το περχόμενο Brexit. Θα ήθελα να μας πείτε λοιπόν ποιοι είναι οι στόχοι σα ό,τι αφορά το μέλλον της Ευρώπης και των νέων με ποιο τρόπο θα καταστήσετε αυτά τα θέματα προτεραιότητά σας. Είπατε και για τα Δυτικά Βαλκάνια ότι χρειάζονται μια σαφή ευρωπαϊκή προοπτική και να έχουν μεταξύ τους συνδεσιμότητα αλλά και μεταξύ τους και με τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να αναφέρω μεταξύ άλλων τη σημασία τη στρατηγική Αδριατική Ιωνίου που μπορεί να είναι μια μεγάλη στρατηγική για την διασύνδεση και τη βελτίωση των περιοχών αυτών. Θα προωθήσετε την εφαρμογή της στρατηγικής Ιωνίου Αδριατικής. Να ζητήσω και συγγνώμη γιατί θα πρέπει να φύγω. Ε, έχω και να παραστώ σε εργασίε μια άλλη επιτροπή. Σε συμβουλίου μου όμω οι συνεργάτε μου θα γράψουν ε, κατά και θα μου μεταφέρουν όλα όσα πείτε. Κύριο Βαν Μίλτεμπουργκ τώρα εκ μέρου τη Άλντε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριο Μίλτον, μου καλωσορίσατε. Κύριε Τριπρόεδρε τη Κυβέρνηση, ήταν πολύ σαφή η παρουσίασή σα και συμφωνώ μαζί σα. Λέτε ότι είναι περίεργο να ξεκινούμε τώρα τη συζήτηση για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ δεν έχουμε συζητήσει πρώτα τι πολιτικέ μα προτεραιότητε. Πού θα βρισκόμαστε το 2030. Ελπίζω εσεί να θέσετε τη συζήτηση αυτή πρώτα να συζητηθούν οι πολιτικέ προτεραιότητε και να ακολουθήσει ο προπολογισμό στο Συμβούλιο ως επόμενο βήμα. Διότι αν ξεκινήσουμε να εστιάζουμε και να συζητούμε ε, απευθεία τα οικονομικά και να μην θέσουμε ε, και να προσπαθήσουμε να βρούμε απαντήσεις στο ερώτημα που θα είναι η Ευρώπη στο μέλλον, θα είναι εσφαλμένη αυτή η προσέγγιση και θα έχουμε χάσει μια μεγάλη ευκαιρία. Καλή προσέγγιση σας λοιπόν. Επίσης, υπογραμμίστε την ανάγκη επενδύσεων στις διεθνωτικές μεταρρυθμίσεις. Έχω μια ερώτηση. Υπάρχουν δύο νομοθετικέ προτάσει για την ενίσχυση των ιδρωτικών μεταρρυθμίσεων του πρόγραμμα υποστήριξη. Είναι μια πρόταση για αύξηση του διαθέσιμου προπολογισμού και μια πρόταση ώστε τα κράτη-μέλη να προετοιμαστούν να προσχωρήσουν ε, στο ευρώ. Πολιτικέ προτεραιότητε για εσά ποιε είναι σε σχέση με τι δύο αυτέ προτάσει, ώστε να σημειωθεί πρόοδο σε αυτό το μέτωπο. Η συνάδελφο Βέστφαλ ήδη τόνισε την ανάγκη να δοθεί προσοχή στο αστικό θεματολόγιο, στην αστική διάσταση των περιφερειακών πολιτικών και των πολιτικών συνεχίσεων. Τα τελευταία δύο χρόνια ξεκινήσαμε αρκετές στρατηγικές εταιρικές σχέσεις, πρώτες τις οποίες έχουν ήδη δώσει ε, σχέδια δράσης. Στο δικό σας πρόγραμμα αναφέρετε κάποια πράγματα. Έχετε συγκεκριμένες ιδέες για αυτές τις στρατικές θεματικές εταιρικές σχέσεις και ο συνάδελφος μου ο Λάμπερντ Φανίστελ Ρόι αυτοπροσκαλείται ε, πάντοτε σε σημαντικές εκδηλώσεις. Ελπίζω να του δώσετε πρόσκληση και να πάνε κι άλλοι τον Ιούνιο σε αυτή την εκδήλωση. Χαίρομαι που προσέχετε την πολιτική συνοχή. Ως συνοχή ε, νομίζω ότι ακριβώς ε, είναι πολύ εύκολο το σλόγγαν σας ισχύσαν τη ενώση. Ευχαριστώ πολύ. Μέρο τη ΓΚΟΕ, τώρα το λόγο έχει ο κύριο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Σομαρζέ, κύριε Πρόεδρε τη Κυβέρνηση. Με χαρά σας ξανασυναντούμε μετά την ε, επίσκεψή μας στη Σόφια, όπου και συγκεκριμένα είδαμε αυτό για το οποίο μας λέει συνέχεια η πρόεδρος της Επιτροπής μας, δηλαδή πόσο η πολιτική συνοχή ε, επηρεάζει ε, την κατάσταση στη Βουλγαρία. Είναι κρίσιμη χρονική στιγμή ε, αυτή. Το δημοσιονομικό μέλλον της Ένωσης είναι αβέβαιο. Κρίσιμη στιγμή και γιατί όλοι μας διερωτώμεθα για το ποιο θα είναι το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Με ικανοποίηση λοιπόν ακούσαμε ότι η Βουλγαρία φίλη χώρα της συνοχής ασκεί την Προεδρία σε αυτήν την πολύ σημαντική χρονική στιγμή. Και βέβαια βασιζόμαστε σε εσά για να προωθήσετε τη συνοχή στο εξάμεινο της Προεδρίας σας. Για να προβάλλετε την προσθεμένη αξία της πολιτικής συνοχής και για να καταπολεμήσετε κάποια στερεότυπα και παροχημένε ιδέε σε ό,τι αφορά την περιφερειακή πολιτική. Και βέβαια κυρίω για να βοηθήσετε στο Συμβούλιο να μην γίνουν ε, χειρότερα τα πράγματα για αυτούς που είναι σε μειονεκτική θέση. Βέβαια θα πρέπει να είμαστε ε, ξεκάθαροι ως προς το ότι υπάρχει η εξής δυσκολία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να τα καταφέρει καλύτερα και να κάνει περισσότερα με λιγότερα μέσα. Είναι μια αντίφαση που πρέπει να ξεπεράσουμε. Και μέσα υπάρχουν για να επικαιρεστεί αυτή τη δυσκολία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προχωρήσει σε ε, δημιουργία νέων ιδιών πόρων. Έκθεση μόντι, να μην σας αναφέρω, τα σχετικά φαντάζομαι τα γνωρίζετε. στο έγγραφο που μας δώσατε. Δεν διάβασα κάτι σχετικό. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε κατά πόσον το θέμα των ιδίων πόρων θα είναι κάτι που θα σας απασχολήσει στη διάρκεια της Προεδρίας σας. Όπως είπατε, το είπε και ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν στη Γαλλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να γίνει ένα συνδικάτο κρίσεων. Αλήθεια είναι αυτό. Ούτε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να θυσιάσει τις κοινωτικέ πολιτικές που κατοχυρώνονται και στις συνθήκες ακριβώς για να ανταποκριθεί στις κρίσεις που έχει να αντιμετωπίσει. Και η πολιτική συνοχής, το λέω και θα το ξαναλέω, είναι η συνοχή, η υποχρέωση κατοχυρωμένη στη συνθήκη. Και αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Επίσης, Άκουσα αυτά που είπατε για τους ελέγχους, πράγματι υπάρχει ανάγκη απλούστευσης. Είμαι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Υπερπολογισμού και μπορώ να σας πω ότι αληθεύει επίσης και το εξή. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες της Ένωσης τίθεται το πρόβλημα της απάτης, της διαφθοράς. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε εσείς αν στο εξάμεινο της Προεδρίας σας θα ε, εντάξετε στις προτεραιότητές σας αυτά τα θέματα. σε ό,τι αφορά το μέλλον τη πολιτική συνοχή, γίνεται πολλή λόγο σήμερα για τη δημιουργία νέων όρων και αιρεσιμοτήτων. Η ομάδα μου, η GUNGL, είναι αντίθετη, το θεωρεί ε, αρχή, ε, στη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Και αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στο να παραμείνουν πιστές οι χώρες της Ένωσης στις ευρωπαϊκές αξίες, στο κράτο δικαίου θα ήθελα λοιπόν και πάνω σε αυτό να ακούσω τις απόψεις σας. Τέλος, γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια σημαντικότατη στρατηγική για τις ε, εξόχως ε, απόκεντρες περιφέρειες. Ανανέωσε τη στρατηγική της για τις περιφέρειες αυτές. Ε, το, η Ολομέλη του Κοινοβουλίου ψήφισε και σχετικό ψήφισμα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα θέλαμε επί της Δικής Προεδρίας να αποφανθεί από αυτή τη στρατηγική και των προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα θέλαμε να είναι και αυτή μια προτεραιότητά σας. Ευχαριστώ. Thank you On Ευχαριστώ. Από τους Πρασίνους, ποιος θα πάρει το λόγο, κύριος Σκάρλετς. Ευχαριστώ. Κύριε Τόντσεφ, καλώς ορίσατε στην Επιτροπή μας και σας ευχαριστώ που προσδίδεται τόσο μεγάλη σημασία στην πολιτική συνοχή στις προτεραιότητές σας. Αυτό είναι πολύ θετικό και μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι και η δική μας ομάδα είναι έτοιμη να υποστηρίξει τη Βουλγαρία στην αποστολή της ε, για να υπερασπίσει το στόχο για την πολιτική συνοχή μετά το 2020 στις συζητήσεις για το μελλοντικό προπολογισμό της Ένωσης. Η Βουλγαρική Προεδρία θα σκεφτόταν την ε, δυνατότητα τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία να δεσμεύονται με την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της περιβαλλοντικής η κυρία ερώτησή μου αφορά το εξή. Έχουμε μια περιοχή που είναι πολύ πλούσια σε βιοπικιλότητα στη Βουλγαρία. Εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να σχεδιαστεί ε, το σχέδιο Αρκαδόμηση στο Κέστεργοξ ε, ε, για να μην ε, βλαπτεί η περιοχή αυτή και να δώσετε τις διαβεβαιώσεις στην Επιτροπή ότι θα γίνει πλήρως σεβαστό το ευρωπαϊκό δίκαιο εμείς θα θέλαμε να μειώσουμε, μα πώς πρέπει να σκεφτούμε πώς θα μειώσουμε την αρνητική αντίκτυπο της κατασκευής του αυτοκίνητου δρόμου. Η κυρία Νταμάτο για το EFTD. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Υπουργό για την παρουσία του εδώ και καλή δουλειά. Διάβασα με ενδιαφέρον το πρόγραμμα εργασίας σας. Αντίθετα σε είδα στο παρελθόν, σε άλλες προεδρίες βλέπω ότι το θέμα της πολιτικής συνοχής είναι παρόν ήδη στις πρώτες σελίδες. Επίσης, σημαίνω την ανακοίνωση για την υλοποίηση μια σημαντική διάσκεψη για την πολιτική συνοχή στον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθο. Το Μάιο και τον Ιούνιο θα έχουμε τις προτάσεις για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο και ο νέο κανονισμός για την πολιτική συνοχή. Ευχόμαστε αυτά τα δύο. Ε, μάλλον ε, θα τα διαχειριστεί η επόμενη Προεδρία, όμως σίγουρα η δική σας Προεδρία θα έχει θεμελιώδη ρόλο στις δύο προτάσεις για το πακέτο για την νομισματική ένωση που παρουσιάστηκε στις 6 Δεκεμβρίου και αφορά το πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και το πιθανό early release ε, του αποθεματικού δράσης. Εγώ θα ήθελα η Προεδρία ε, ουσιαστικά να μην ικανοποιήσει τις ε, πολύ επικίνδυνες προτάσεις της Κομισιόν αλλά να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο και με αυτή την Επιτροπή. Μεταξύ των προτεραιοτήτων ε, βλέπω ότι βρίσκεται και ευχή για μια σταθερή, αλληλέγγυη, ισχυρή Ευρώπη και επιμένω σε αυτή την πτυχή στο βαθμό που ξέρουμε ότι ένα μέρος των διαφορετικών επενδυτικών ταμείων χρησιμοποιούνται και το ίδιο θα γίνει και στο μέλλον για την καταπολέμηση της μετανάστευσης. Στη Βουλγαρία έχουμε κάποιες περιοχές που καθυστερούν στην ανάπτυξη και το ίδιο ισχύει και στη χώρα μου. Όλοι γνωρίζουμε ότι ιδίως στην Ιταλία και στην Ελλάδα κάποιες περιφέρειες δέχονται μεγάλες μεταναστευτικές πιέσεις και θα αναγκαστούν να χρησιμοποιήσουν την συσφορά τα διαρθρωτικά ταμεία για να καταπολεμήσουν ή να υπερασπίσουν την επικράτεια δουλειά για να αντιμετωπίσουν καλύτερα την μεταναστευτική πρόκληση. Όμως η συγκεκριμένη εφαρμογή της αρχής της ελληνικής και της ίση κατανομής των μεταναστών σε όλα τα κράτη-μέλη δεν είναι σήμερα κάτι που έχει υλοποιηθεί. Δεδομένου ότι η αρχή του fair burden sharing ε, ε, ουσιαστικά δεν ελαμβάνεται στο Συμβούλιο, θα ήθελα να αφιστήσω την προσοχή σας σε αυτή την προβληματική και εύχομαι οι διαπραγματεύσεις, οι μελλοντικές στο θέμα της συνοχής να λάβουν υπόψη και αυτή την αρχή και για να λάβετε υπόψη και την ε, εφαρμογή της αρχής της ελληνικής που δεν μπορεί να μένει σε απλή διακήρυξη απόψεων αλλά θα πρέπει να μεταφραστεί σε συγκεκριμένες πράξεις ε, λειτουργικές έτσι όπως έχει συλληφθεί η Ευρώπη από τους ιδρυτές πατέρες μιλάμε ε, για ενότητα στην ποικιλομορφία και θα έλεγα και στις δύσκολες στιγμές. Ευχαριστώ πολύ. Έχω κάποιους ακόμη ομιλητές στον κατάλογο και θα πρότεινα να συνεχίσουμε με τις ερωτήσεις και κατόπιν θα δώσουμε το λόγο στον Υπουργό για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις μαζί. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Παπαδημούλη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω τον Αντιπρόεδρο της Βουλευτικής Κυβέρνησης, τον κύριο Τόντσεφ, και να πω ότι άκουσα με ικανοποίηση όσα μας είπε για την ε, πολιτική συνοχής και πώς την βλέπει η Βουλγαρική Προεδρία. Γιατί και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε την ίδια ακριβώς άποψη ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να μην αποδυναμωθεί γιατί έχει αποδείξει διαχρονικά την αποτελεσματικότητά της και την αναγκαιότητά της πολύ περισσότερο που τα τελευταία χρόνια έχουμε μια επικίνδυνη αύξηση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των κοινωνικών και των περιφερειακών ανισοτήτων. Άρα χρειαζόμαστε και ενίσχυση, θα σας έλεγα, της πολιτικής συνοχής. Γι' αυτό ε, η ερώτησή μου είναι, πρώτον, πώς βλέπετε ως Βουλγαρική Προεδρία την ιδέα να εξευρεθούν και νέοι πόροι στο νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, αξιοποιώντας και ιδέες της Επιτροπής Μόντι. Και το δεύτερο, πριν από λίγες εβδομάδες υπογράφηκε μία σημαντική κατά τη γνώμη μου συμφωνία μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Βούλγαρου Πρωθυπουργού, Τσίπρα Μπορίσοφ, για τη δημιουργία κοινών επενδυτικών σχεδίων που να αναβαθμίζουν τους σιδηροδρόμους, τα δίκτυα, τα λιμάνια της περιοχής Νομίζω ότι αυτό είναι μια σημαντική ενίσχυση της περιφερειακής πολιτικής. Και το ερώτημα είναι αν προσβλέπετε ως Βουλγαρική Προεδρία την ενίσχυση, όχι μόνο με ιδιωτικούς πόρους, αλλά και με κοινοτικούς πόρους αυτών των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων. Σας ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Πυρίνσκι. Ε, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ε, αξιότιμε αντιπρόεδρε της κυβέρνησης. Ε, ε, θα ήθελα να ενώσω και εγώ τη φωνή μου με τα συγχαρητήρια των συναδέλφων για τις προτεραιότητες που μας παρουσιάσετε ιδιαίτερα τις προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής. Πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, τονίσατε το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει ε, και τις διαφορές ανάμεσα σε φτωχές και πλούσιες χώρες και φτωχές και πλούσιες περιφέρειες. Αυτό το πρόβλημα είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τη μελλοντική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν θέλουμε να είναι μια σταθερή ε, ένωση και μια κοινότητα αναπτυσσόμενη συνεχώς και όχι ένας μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων. Ε, σε σχέση με όλα αυτά ε, έχουμε την επικείμενη συζήτηση για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Εσείς τι πιστεύετε, είναι απαραίτητο να εστιάσουμε στο να κατανοήσουμε ότι είναι το βασικό εργαλείο για επενδύσεις αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική συνοχής. Γιατί εμείς μιλούμε ε, για αναδιάταξη, ανακατάταξη των προτεραιοτήτων ε, των επενδυτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να τα ξαναδούμε αυτά από την αρχή. Και κάτι άλλο που ε, αναφέρεται και στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η νέα στρατηγική για την εκβιομηχάνηση στην Ευρώπη. Εκεί ε, εστιάζουν και εκεί δίνουν έμφαση πλέον και όλα αυτά συμβαδίζουν ε, με τον πρωτοπόρο ρόλο που θέλει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη νέα βιομηχανική εποχή. Για να μην ακρηγορήσω, θέλω απλώ να αναφέρω κάτι που είπε στην συνάδελφο βέσφαλ προηγουμένως. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα ε, κατά πλειοψηφία ε, και το υπερψήφισαν πολλοί συνάδελφοι από πολλέ πολιτικέ ομάδε. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εποφεληθεί ε, από αυτή την έκθεση του Κοινοβουλίου ε, για να τη μεταφράσει σε πρακτικές πολιτικές. Σε ό,τι αφορά τώρα το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, είναι προφανές ότι αυτό που κυριαρχεί εκεί ή θα κυριαρχήσει είναι αυτό που και αναφέρετε και εσείς, ότι πρέπει να επιτύχουμε περισσότερα με λιγότερα μέσα ενδεχομένως. Κάποιοι συνάδελφοι σωστά πρότειναν να κατευθυνθεί η συζήτηση ε, προς τα έσοδα και τους ιδίους πόρους της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μελλοντική της χρηματοδότηση. Επίσης αναφερθήκατε σε μια επανάσταση που χρειάζεται να γίνει. Πραγματικά έχετε δίκιο. Ε, χρειάζεται βαθιά αλλαγή νοοτροπίας και σκέψης για τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχουν διάφορες χώρες στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πολιτική της δίκαιης απόδοσης αυτό που λένε στα γαλλικά «juste retour» ότι θέλω να πάρω πίσω όσα δίνω είναι μια ιδέα που μπλοκάρει τα πράγματα και δεν βοηθάει. Ο Επίτροπος Τιγκέρ προσπαθεί να αλλάξει αυτή την οτροπία και να αλλάξουν και τα Ε, πράγματα ως προς τους ιδίους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από πού θα αντιληθούν αυτά τα κονδύλια. Από το φόρο χρηματοπιστωτικών ε, συναλλαγών ή το τέλος ε, χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Ανησυχούν πολύ εδώ στο Κοινοβούλιο για το μέλλον αυτής της πολιτικής και για τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες. Εκεί λοιπόν χρειάζεται επανάσταση, αλλαγή νοοτροπίας, αλλαγή τακτικής για να αποζημιωθούν ή να αντισταθμιστούν οι απώλειες από το Brexit στα δημοσιονομικά. Σε ό,τι αφορά τώρα την εφαρμογή των πολιτικών, ανέφερε ο κ. Ρόι ότι υπάρχουν διάφορες ιδέες ε, συνδυασμός διαφόρων ταμείων, εξαίρεση κάποιων ταμείων από την πολιτική συνοχής. Κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό να μην χαλάσουμε κάτι που λειτουργεί σωστά αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν είναι, έτσι λέει η λογική. Παρακαλώ, πείτε μας την άποψή σας. Θεωρείται σκόπιμο να συνενωθούν διάφορα χρηματοδοτικά μέσα που ε, αυτή τη στιγμή είναι σε διαφορετικά προγράμματα. Στο πρόγραμμα ε, συνδέοντας την Ευρώπη, ας πούμε, ή άλλα. Μαζί με το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων γίνονται διάφορες προτάσεις, ακούγονται διάφορες ιδέες, αλλά χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή εδώ και στάθμιση των διαφόρων παραγόντων. Υπάρχει ένας κίνδυνος το ανέφερε και ο κύριος Βανίστερόι. Μήπως επικρατήσει κάποια σύγχυση ε, όταν μπαίνουν διάφορες πολιτικές και διάφορες πηγές στο ίδιο τσουφοχάλι. Και θέλω να σας αναφέρω μια ανησυχητική στατιστική που διάβασα. 20% είναι οι πληρωμές φέτος που διανύουμε τον τέταρτο χρόνο της προγραμματικής περίοδου ενώ το αντίστοιχο έτος προηγούμενης περίοδου ήταν 40% η απορρόφηση των κονδυλίων πάντα στο τέταρτο έτος. Αυτό τι σημαίνει ότι η εξάντε αιρεσιμότητα και οι διάφοροι κανόνες και όροι που έχουν μπει δυσκολεύουν τα πράγματα. Και θα πρέπει να το δει αυτό το Συμβούλιο, να συνεχιστεί αυτή η πρακτική. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ φλέγων. Θα πάει έτσι και η επόμενη προγραμματική περίοδος. Μήπως πρέπει να σταματήσει αυτό. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε να μιλήσω και ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Mm, Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θέλω να σας ευχηθώ ε, κάθε επιτυχία στην ε, Βουλγαρική ε, Προεδρία. Έρχομαι από την Τσεχία. Έχουμε παρόμοια προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Ε, πολλά είναι τα ζητήματα, δεν θα τα επαναλάβω. Τα είπαν προελίσσαντε συναδελφοί μου. Μιλήσατε όμω ε, στην προσφώνησή σα για κάποια ζητήματα που τα θεωρώ σημαντικά. Το πρώτο αφορά τη διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημά μου είναι, η Βουλγαρική Προεδρία πώ θα υποστηρίξει τη διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλήσατε για τα Βαλκάνια και το εκτίμησε όλος ιδιαιτέρως. Πιο συγκεκριμένα όμως, πώς θα πείσετε τα κρατη που είναι άκρος επιφυλακτικά. Η δική μου θέση και η θέση της χώρας μου είναι η υποστήριξη της διεύρυνσης. Εσείς απαριθμίσατε τους λόγους ε, ε, που έχουν να κάνουν με την περιοχή αυτή. Ότι πρόσωπο του Κοινοβουλίου δεν είναι εδώ τέλος πάντων. Ε, στην παρέμβαση σας είπατε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα με λιγότερα. Αν δεν έχουμε στην Ένωση όμως νέους πόρους, από πού θα κόψουμε και τι ε, θα περικόψουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ε, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρόπε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω και εγώ τον αντιπρόεδρο της αυλγαρικής κυβέρνησης. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Χαίρομαι ιδιαίτερω με αυτά που άκουσα να λέτε σε ό,τι αφορά τι προτεραιότητε σας. Είναι πολύ θετικό ότι έχουμε κοινέ προτεραιότητες. Βέβαια το σημαντικότερο είναι εμείς να συμφωνήσουμε και επί της εφαρμογής των προτεραιότητων. Πώ από κοινού θα τι εφαρμόσουμε. Το Brexit είναι σίγουρα ένα ζήτημα το οποίο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ε, τομέων ε, και αφορά τον υπερπολισμό. Εσείς που κλείνετε, ποια είναι η άποψή σας. Πρέπει να συμφιλεφούμε την ιδέα ότι στο μέλλον θα έχουμε λιγότερους πόρους, άρα θα πρέπει να δαπανίσουμε και λιγότερα χρήματα ή μήπως θα έπρεπε τα κράτη-μέλη αντίθετα να εξετάσουν το δεχόμενο να αυξήσουν τη συνεισφορά τους και σε ό,τι αφορά τρίτη προτεραιότητα που αναφέρατε, μιλήσατε για το ενδεχόμενο να σκεφτούμε ε, και άλλους ίδιους πόρους. Ποια είναι η επιλογή που προτιμάτε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική συνοχή, ε, ή τέλο με τη βοήθεια τη πολιτική συνοχή, Ε, θα έχουμε αντιμετωπίσουμε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών. Μπορεί και να είναι πολλαπλάσιες ε, των σημερινών διαφορές και έχουμε και διαφορές μεταξύ αστικών και ευρωτικών περιοχών. Κατά την άποψή σας στο μέλλον θα χρειαστούμε ένα μηχανισμό που θα υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να μειώσουν την ψαλίδα μεταξύ των ε, πιο πλούσιων και των πιο φτωχών περιφερειών τους. και κάπως να προς, ε, ε, εξομοιωθεί το βιωτικό επίπεδο μεταξύ των κρατών μελών. Αν υπάρχει αυτό το μεγάλο χάσμα και στη συνέχεια αυτό θα δημιουργήσει δυσαρέσκεια και θα αυξήσει τα μεταναστευτικά ρεύματα. Το ερώτημα για την πολιτική συνοχή είναι ο κόσμος καταλαβαίνει η Δήμη, η διοίκηση συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τον προπολογισμό. Η κοινωνία των πολιτών και άλλοι φορείς συμμετέχουν τελικά. Αυτό είναι προϋπόθεση. Πρέπει να συμμετέχουν στις αποφάσεις που τους αφορούν όλοι αυτοί οι φορείς. Και οι περιφέρειες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία λήψη αποφάσεων γιατί τους αφορούν αυτές οι αποφάσεις. Και έτσι θα έχουμε περισσότερη απασχόληση και μεγαλύτερη ανάπτυξη. Υπάρχει ένα άλλο κακό που δεν το έχουμε ε, ακόμη αντιμετωπίσει. Ότι οι λίγες πλούσιες περιφέρειες ε, γεννούν πολύ πλούτο, ο οποίο όμως ε, πηγαίνει πάλι σε πλούσιες περιφέρειες. Ε, υπάρχει επίσης απώλεια φορολογικών εσόδων πολλές φορές. Δεν πηγαίνει ο πλούτος στις περιφέρειες. Πρέπει να βρεθούν λύσεις. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και αυτό το πράγμα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ και τέλος να σας πω ότι από τις αποφάσεις μας θα εξαρτηθεί το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Πιθανότατα θα έπρεπε να μιλήσω βουλγαρικά. Όμως ακούγοντας τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ε, σκέφτηκα ότι μπορεί να ακούγεται ε, κάτι σαν σενάριο ταινία του Χόλιγουντ ε, ή στρατιωτικός όρος όμως ευρωπαϊκός προπολογισμό. Ε, ε, και η πολιτική συνοχή δεν θα έπρεπε να αφήνει τους ανθρώπους ε, πίσω, Εκτό θα έπρεπε να μπορούμε να απευθυνθούμε σε όλους παντού και πάντοτε. Ένα συνάδελφό μου μου είπε πρόσφατα ότι η βουλγαρική προεδρία μπορεί να θεωρηθεί κατάρα αν σκεφτούμε την χρονική στιγμή της ανάληψης της Προεδρίας. Υπάρχουν τόσο δύσκολα και κατεπήγοντα ζητήματα και κάποια προβλήματα φαίνονται ανεπίλητα. Είναι αυτό η ιδιαίτερη ευθύνη της Βουλγαρικής Προεδρίας. Και θα πρέπει να φέρετε αυτό το άχθος και να ανεβείτε τις βουνοκορφές. Εγώ βλέπω εδώ ένα εμπόδιο το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο το οποίο θα συζητηθεί και κατόπιν το προτινόμενο νέο κανονισμό και η εφαρμογή του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο ισχυρή όσο το πιο αδύναμο κράτος μέλος. Ακούω φωνές που υποστηρίζουν την πολιτική συνοχή και άλλες που δεν την υποστηρίζουν. Κατά την άποψή μου υπάρχουν δύο κατηγορίες χωρών. Χώρες που ανοιχτά υποστηρίζουν την πολιτική συνοχή και μια άλλη ομάδα χώρες που δεν ε, το παραδέχονται ότι την υποστηρίζουν δημοσίως. Γιατί η πολιτική συνοχής ωφελεί περισσότερους από τις χώρες δικαιούχος. Όταν ανοίγουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για επενδύσεις δεν υποστηρίζουμε απλώ ε, τα βουλγαρικά ή τα ρουμανικά έργα. Έτσι λοιπόν η χρηματοδότηση των μεγαλύτερων έργων είναι ζωτικού ενδιαφέροντο. Υπάρχουν κάποιε ακραίε απόψει ότι η πολιτική συνοχή ε, συμπεριλαμβανομένων και των άμεσων πληρωμών ε, θα πρέπει να περιοριστεί και ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι εθνικοί συντελεστές χρηματοδότηση. Εγώ δεν υποστηρίζω μια τέτοια ιδέα. Υπάρχουν κάποιες τρίτες χώρες ε, που θα ήθελαν να επενδύσουν ε, σε κάποια σημαντικά έργα υποδομής. Ε, βέβαια πρόκειται για αλλοδοπείς εταιρείε και φέρουν και τα δικά τους ξένα συμφέροντα και τους δικούς τους αλλοδαπούς όρους. Και επιπροσθέτως έχουμε και τον Brexit. έχουμε ένα κράτος μέλος που πρόκειται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν υπολογίσουμε τη συνεισφορά της και το μερίδιό της στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τότε το ποσό γίνεται τεράστιο, γίνεται υπέρογκο. Μπορεί να φτάνει και τα 100 δισεκατομμύρια. Και είναι πολύ σημαντική απόφαση για το πώς θα καλυφθεί αυτό το κενό που θα προκύψει. Θα ήθελα να μου απαντήσετε στην ερώτηση αυτή λοιπόν. Υπάρχει μια γερμανική λέξη, ώρας Waffenrute. Ε, υπάρχουν ε, άνθρωποι που συμφωνούν με τις ιδέες σας. Πρόκειται για το αδερφού στα όπλα. Και έχετε εδώ αδερφού στα όπλα, σε αυτή την αίθουσα. Θα βρείτε υποστηρικτές. Και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Νοβάκοβ. Και τώρα έχει ώρα, έρθει η ώρα να απαντήσετε. Ε, ακούσατε τις ε, απόψεις των συναδέλφων. Ε, θα ήθελα να πω και εγώ δύο λόγια ως πρόεδρος ε, της παρούσης Επιτροπής. Τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες και έχει αποκομίσει και κάποια εμπειρία. Και θα ήταν όμως τώρα χρήσιμο και σωστό τώρα που παίρνουμε τις αποφάσεις για το μέλλον της πολιτικής συνοχής να λάβουμε υπόψη μας κάποιες εκθέσεις που έχουμε εμείς εδώ ιδίας πρωτοβουλία, για το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, για την κυκλική οικονομία, για την πολιτική συνοχής. Έχουμε εκθέσεις ε, για την ανάπτυξη ε, την περιφερειακή, την εδαφική, την αστική. Όλες λοιπόν αυτές οι εκθέσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της φαρούσης αλλά και της μελλοντική πολιτικής συνοχής. Έχουμε εργαστεί επί πολλών ε, νομοθετικών θεμάτων που ε, προεξοφλούν τις μελλοντικές τάσεις της πολιτικής συνοχής όπως είναι η δημοσιονομική ευελιξία. Έχουμε ακούσει πολλές συζητήσεις, έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις για την υποστήριξη που πρέπει να δοθεί στα κράτη-μέλη που πλήττονται από θεομηνίες. Έχουμε συζητήσει και για συγκεκριμένες χώρες, την Ελλάδα, την Κύπρο, επίσης το πακέτο Omnibus το πρώτο που οδήγησε στην ουσιαστική απλούστευση των διαδικασιών και τη βελτίωση της προβολής της πολιτικής συνοχής. Έτσι δόθηκε ευκαιρία στους δικαιούχους να χρησιμοποιούν τα κονδύλια με ευελιξία, καθώς επίσης και να χρησιμοποιούνται τα κονδύλια της συνοχής για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και πιέσεων. Η κυκλική οικονομία είναι επίσης σημαντική. Η έβδομη έκθεση ε, συνοχής πρόκειται να δημοσιευτεί προσεχώς. Και η Επιτροπή μας θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει ε, τα θέματα αυτά και να πάρει σημαντικές αποφάσεις. Είχαμε πολλές συνεδριάσεις, συναντήσεις με συναδέλφους, με την Επιτροπή των Περιφερειών, με πολλές ευρωπαϊκές ενώσεις και οργανώσεις. Γιατί τα απαριθμώ όλα αυτά, διότι είμαι πεπισμένη ότι τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης θα πρέπει να συμμετέχουν σε βασικές προτεραιότητες και βασικές πρωτοβουλίες μάλλον ε, της Βουλγαρικής Προεδρίας ε, στη συνοχή μπορούμε να έχουμε πολύτιμη πραγματικά συνεισφορά. Και συμφωνώ με όλους τους συναδέλφους που υποστήριξαν πλήρως τις βουλγαρικές προτεραιότητες ε, της πολιτικής συνοχής. Ολοκληρώνω εδώ και δίνω το λόγο στον Υπουργό για να απαντήσει. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, απαντώ. Ήταν πολύ καλά τα ερωτήματα που θέσατε πραγματικά πάρα πολύ ε, καλά ερωτήματα γιατί μας δίνουν τη βάση για να έχουμε μη ειλικρινή ε, ανοιχτή συζήτηση. Δεν καλό να αναμασάμε βέβαια τα ίδια και τα ίδια και νομίζω ότι η πρώτη μας συνάντηση δίνει το πολύ καλό παράδειγμα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω ότι εσείς ε, ως το πιο αναλυτικά. Αν όμως δεν μπω σε λεπτομέρειες, ε, θα σας ε, γλιτώσω και από το να μείνω μέχρι τα μεσάνυχτα εδώ. Για το ρόλο του Κοινοβουλίου της Κομισιόν, για το πώς βλέπουμε τη συνεργασία μας, κάποια λόγια. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας αποκαλώ συναδέλφος γιατί επί μισή μήνες ήμουν μέλος της κοινοβουλευτικής αυτής επιτροπής και κάποιους από εσάς σας γνωρίζω από τότε. Δεν έχει σημασία για το κατά πόσον μιλάμε για εθνικά κοινοβούλια ή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι αυτό μόνο ένας αντιπροσωπευτικός οργανισμός. Είναι και θα πρέπει να είναι ένα εργαστήρι ιδεών που θα μας δώσει νέες ιδέες, νέες προκλήσεις, κάτι το οποίο χρειαζόμαστε πάρα πολύ σήμερα. Θα χαρώ πολύ λοιπόν να σας δω και ανεπισήμως, αλλά και σε οποιαδήποτε εκδήλωση για τις συζητήσεις που θα έχουμε και τις εκδηλώσεις. Δεύτερον, με βάση την εμπειρία μου στο ό,τι αφορά το προπολογισμό και την πολιτική συνοχή, η εντύπωση που αποκόμισα είναι ότι προτείνουμε να υπερασπιζόμαστε συνεχώς την πολιτική συνοχή. Λάθος τα λέμε. Πρέπει να αναδιατυπώσουμε και να ε, αναδιοργανώσουμε την όλη συζήτηση. Δεν θα πρέπει να υπερασπιζόμαστε την πολιτική συνοχή. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θέλει να την καταστρέψει. Το ζήτημα είναι πώς θα τη βελτιώσουμε την πολιτική συνοχή. Θα ήθελα να εκφράσω την ε, πεποίθησή μου ότι η όλη συζήτηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα δείξει ε, τι εμπιστοσύνη έχουν σε αυτούς μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μιλάμε για την πολιτική συνοχή, κάποιοι τείνουν ε, να θεωρήσουν ε, ότι έχει να κάνει μόνο με λογιστικά πρότυπα, έσοδα, δαπάνες ή σε φιλανθρωπία. Καμία σχέση. Πρόκειται για ένα επενδυτικό σχέδιο που ξεκίνησε από το να καλύψει κάποια κενά της αγοράς, αλλά έχει προσθέμενη αξία πολύ σημαντικότερη. Επενδύσεις στην Ευρώπη, επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ είμαστε μια λέσχη ανθρώπων που ανταλλάσσουμε ιδέες. Θα πρέπει να είμαστε ένας κλειστός κύκλος, μια κλειστή κοινότητα που αμφαλοσκοπεί. Θα πρέπει όλοι να έχουν ε, το λόγο τους και όλοι να ακούγονται. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτικό χρέος. Εγώ θα αξιοποιήσω κάθε δυνατότητα και οποιοδήποτε άλλο συμβάν ε, και οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση συνέδρια, διασκέψεις, ε, ψηλού επίπεδου συναντήσεις ε, για να έχουμε συζητήσεις στο άλλο δυνατό επίπεδο. Εκεί θα διερευνήσουμε τις ανάγκες, θα ανταλλάξουμε ιδέες, θα κάνουμε την προκαταρκτική μας ανάλυση. Θα δούμε ποιες είναι οι απόψεις των πιο ε, σημαντικών πρωταγωνιστών της όλης αυτής διαδικασίας και ιδίως τι προοπτικές υπάρχουν για την περίοδο μετά το 2020. Πρέπει να σας πω ότι από την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο παρατηρώ κάτι σημαντικό. Δεν είμαστε σε πολύ καλή συγκυρία. και από την περίοδο 2007-2013. Αντί να έχουμε οικονομική άνθηση και πρόοδο, αντιμετωπίσαμε την οικονομική κρίση, την ύφεση. Και ο προγραμματισμός για την επόμενη περίοδο έγινε με αυτές τις παραμέτρους. εκεί που η προηγούμενη περίοδος είχε ε, σχεδιαστεί με βάση την ευημερία που δεν έγινε πράξη, αυτή η περίοδος έχει σχεδιαστεί με βάση μια κρίση που ελπίζουμε να μην μείνει έτσι και να Δεν πρέπει λοιπόν να είμαστε ε, όμοιροι αυτής της εξάρτησης από τις συγκυρίες. Ένα άλλο θέμα ε, πολύ σημαντικό αφορά τον κοινωνικό πυλώνα. Και είναι άκρος επίκαιρο το θέμα αυτό. Διότι τελικά το ανθρώπινο κεφάλαιο, η ανεργία, η απασχόληση, τα δημογραφικά ζητήματα είναι στο μυαλό όλων. Το κοινωνικό ταμείο, τα μέτρα, ε, τα κοινωνικά είναι πολύ σημαντικά. Και ναι, παρατηρούμε και παρακολουθούμε τα μηνύματα και τα σημάδια των καιρών. Έχω να σας πω το εξής. Θεωρώ ότι e Έχουμε τους πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Δεν υπάρχουν ε, μόνο αυτοί βέβαια οι πόροι. Αλλά είναι σημαντικοί. Θέλουμε επίσης ολοκληρωμένες πολιτικές Δεν μπορούμε να κατανέμουμε τα προβλήματα ανάλογα με τους πόρους. Δηλαδή να πούμε ότι το τάδε πρόβλημα θα λυθεί από τα κονδύλια του Ταμείου Συνοχή, το δεύτερο πρόβλημα από το επενδυτικό και δεν ξέρω από τι. Θα πρέπει να τα δούμε ταυτόχρονα και ολιστικά. Είναι πρόκληση και το αντιλαμβάνομαι. Να έχουμε εργαλεία κατάλληλα προσαρμοσμένα για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε εξατομικευμένα τα προβλήματα. Και δεν είναι εύκολο να προέλθει ε, χρηματοδότηση από ένα ταμείο για ένα πρόβλημα και χρηματοδότηση από ένα άλλο ταμείο για ένα άλλο. Και, για μένα, Γνωρίζω ότι επί Βουλγαρικής Προεδρίας δεν έχουμε κάποια ειδικά δικαιώματα, έχουμε όμως σίγουρα υποχρεώσεις ειδικέ. Σίγουρα τα κοινωνικά ζητήματα θα αποτελέσουν ένα απόσπαστο κομμάτι της πολιτικής συνοχής. Γιατί είναι πολύ σημαντικό τμήμα της πολιτικής συνοχής ούτως ή άλλως. Η επιβίωση της πολιτικής συνοχής δεν πρέπει να αποτελεί αυτό σκοπό. Πρέπει να τα καταφέρουμε καλύτερα σε πολλούς τομείς. Πρόκειται για μια προσέγγιση που βασίζεται στην αλληλεγγύη, αλλά όχι στη φιλανθρωπία, παραλαμβάνω. Και κανείς δεν πρέπει να πει ότι εμείς είμαστε ένα νέο κράτος μέλος, είμαστε μια φτωχή χώρα. Βοηθήστε μας λοιπόν, γιατί είναι καθήκον σας όχι. Ε, αυτό το επιχείρημα να ξεχαστεί. Όλοι μας θέλουμε και πρέπει να γίνουμε πιο πλούσιοι. Όλοι μας. Βάσει πολιτική συνοχής. Και η πολιτική συνοχή θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά την άποψη όλες τις περιφέρειες της τη Να μην ξεχνάμε ότι δεν πρόκειται για μια πολιτική μόνο για τις απόκεντρε ή για τις πιο φτωχές περιφέρειες ή αυτές που χρειάζονται πιο ταχεία συνοχή. Πρέπει να στοχεύσουμε υψηλότερα στην καινοτομία, να δώσουμε έμφαση στη γνώση, στην κοινωνική ένταξη, στην παιδεία. Ακόμα και στις πιο πλούσιες χώρες της Ένωσης. Αυτά είναι χαρακτηριστικά θέματα. Στο αστικό θεματολόγιο αναφερθήκα το ορισμένο. Είναι πράγματι. Είναι πολύ σαν τη Φραγκφούρτη, για παράδειγμα. Όπως παλιότερα το Λονδίνο πριν το Brexit που δεν έχει γίνει ακόμη είναι από τις πλουσιότερες πόλεις του κόσμου. Έχουμε καταφέρει όμως να μην περιοθεοποιήσουμε αυτούς που χρειάζονται βοήθεια εκεί. Πώς θα πείσουμε τους πολίτες ότι είναι καλή πολιτική συνοχής εάν μόνο σε κάποιες χώρες εφαρμόζεται και όχι σε άλλες. Ανταυτού εγώ νομίζω ότι πρέπει να είναι μια πανευρωπαϊκή πολιτική ως, αν θέλετε, παιδαγωγική άσκηση. Ένα άλλο ερώτημα, φως την ευελιξία. Πολύ καλό ερώτημα. Όπως είπα, σχεδιάζουμε κάποια μέτρα σε έναν κύκλο, τα οποία εφαρμόζονται σε έναν άλλο κύκλο. Και μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα τελικά. Άρα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι. Η ευελιξία όμως έχει τα ωριά της. Μπορεί να θέλουμε να δαπανίσουμε κάποια χρήματα για την ε, τάδε κρίση, τη δίνα κρίση ή άλλε προκλήσει. Αν το κάνουμε αυτό, κινδυνεύουμε να χάσουμε τον αρχικό στόχο της πολιτικής συνοχής. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται καν να σα εξηγήσω. Ποιο ήταν ο αρχικό στόχος τη πολιτικής συνοχής. Που ήταν η άρση των ανισορροπιών Φυσικά και πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να αντιμετωπίζουμε τις τρέχουσες προκλήσεις και κρίσεις, αλλά να μην μας παρασύρει αυτή η ιδέα. Γιατί κάποια προβλήματα χρειάζονται δεκαετίες ολόκληρες για να επιληθούν. Μίλησα για επανάσταση. Μ' αρέσει η λέξη επανάσταση. Επίσης τι μπορούμε να κάνουμε για την απλούστευση. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Όλες τις αντλούμε από την εμπειρία μας. Ψηφιοποίηση, το πρώτο. Το έχουμε πράξει. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα εξαφανιστεί το χαρτί. Αυτό είναι καλό. Και το καλό είναι ότι θα έχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα στις συναλλαγές ή τις ε, πράξεις. Θα υπάρχει ίχνος, αποτύπωμα και άρα έλεγχος όλων αυτών των πράξεων και συναλλαγών. Έχουμε επίσης την ανάγκη να αναπτύξουμε τυποποιημένα λογιστικά ε, πρότυπα για τα έσοδα και τις δαπάνες. Και έχουμε εμπειρία, δεν ναι, βλέπω το λόγο γιατί δεν θα πρέπει να βάλουμε τον πύχη ψηλότερα στο ευρωπαϊκό επίπεδο για να έχουμε παραδείγματο χάρη τυποποιημένα έγγραφα και στις δημόσιες συμβάσεις, τους σχετικούς διαγωνισμούς. Υπάρχει τυποποιημένη, ε, τυποποιημένα έγγραφα, υπάρχουν σε πολλές περιπτώσεις και αν έχουμε λοιπόν στις δημόσιες προμήθειες τυποποιημένα έγγραφα θα υπάρξει και μεγαλύτερη διαφάνεια. Έρχομαι στο μέλλον των νέων. Θα περιμένετε ένα κλισέ από μένα, φαντάζομαι, ή να επαναλάβω τα γνωστά προβλήματα. Ανεργία των νέων, που είναι ένα σοβαρό πρόβλημα, ιδίω ορισμένα κράτη-μέλη, τα κράτη-μέλη του Νότου. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να αναλύσουμε πολύ πιο επακριβώς τα αίτια της ε, ανεργίας των νέων. Πού οφείλεται, στις αγορές, στην κοινωνική συμπεριφορά, στις συμπεριφοριστικές προκλήσεις. Πρέπει να εντοπίσουμε τα προβλήματα των νέων και τι καλύτερος τρόπος από το να συμμετέχουν οι νέοι στη διαδικασία αυτή. δεν μου αρέσει όταν μια ομάδα μιλά για μια άλλη χωρίς αυτή η ομάδα να συμμετέχει. Ε, είμαι επιφυλακτικός απέναντι στα πορίσματα που θα βγουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι μακροπεριφέρειε και μικροπεριφερειακές στρατηγικέ, νομίζω ότι είναι μια χρήσιμη προσέγγιση. Και αφορά και τα Δυτικά Βαλκάνια. που ανήκουν στην ε, περιφέρεια του Δούναβη, άρα συμμετέχουν στη στρατηγική του Δούναβη και σε άλλες περιφέρειες που καλύπτονται με μακροοικονομικές στρατηγικές. Και έχει αλλάξει η εμπειρία τους και η νοοτροπία τους λόγω αυτής της συμμετοχής. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και γενικά αλλά και ειδικά Έχουμε κάποιες αλλαγές με τον νέο κανονισμό. Εγώ μπορώ να σας πω ότι ο στόχος μας είναι να πετύχουμε τη συνένεση. Δεν θέλω όμως αυτό να φανεί ότι αποφεύγω να απαντήσω συγκεκριμένα. Γι' αυτό και θα σας απαντήσω συγκεκριμένα. Πρέπει σε όλη την Ευρώπη οι μεταρρυθμίσεις να γίνονται με τον ίδιο ρυθμό, ναι, είναι η απάντηση. Όπως όταν μιλάμε για τη συνοχή και τη σύγκληση. Υπάρχουν κάποιες χώρες πιο σύγχρονες, πιο προηγμένες. Και αυτό είναι... Τι πρόβλημα υπάρχει, πού υπάρχουν οι ελλείψεις, τι πρέπει να αλλάξει. υπάρχει πολιτική βούληση και το στένος για να γίνει κάτι τέτοιο. Όλες αυτές οι προκλήσεις είναι υπαρκτές. Ο σχεδιασμός έγινε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πιστεύω. Πήραμε ως παράδειγμα το καλύτερο. Αλλά πρέπει να υπάρχει και το απαραίτητο πολιτικό στένος για να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις γιατί αυτές οι βέλτιστες πρακτικές δεν είναι κάτι μυστικό, είναι γνωστές. Σίγουρα υπάρχουν εθνικέ ιδιαιτερότητες στον τομέα της δημόσιας διοίκησης, της υγείας, ε, της παιδείας, της αγορά εργασίας, την οικονομική διακυβέρνηση. Οι τοπικοί πολιτικοί γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, ε, απάτη και διαφθορά. Ελπίζω να μην ε, θεωρήσατε αυτά που είπα για ριζική απλούστευση ως μία πρόφαση ε, ανοχής της διαφθοράς και της απάτης. Όχι, μηδενική ανοχή. Η ψηφιοποίηση επιτρέπει πλήρη έλεγχο ε, σε πραγματικό χρόνο. Αυτή είναι η απόφαση και αυτή είναι η λύση. Ο ευφυής έλεγχος. Προσπαθούμε να είμαστε συγκεκριμένοι, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε και χρήσιμοι. Ε, και προσπαθώ να απαντήσω και εντό του χρόνου που έχουμε ακρίβεια. Χρειαζόμαστε βιομηχανία με μεγαλύτερη ε, προστιθέμενη αξία. Γι' αυτό χρειάζονται επενδύσεις σε τεχνογνωσία, ε, στην ανάπτυξη, στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στην καινοτομία. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί σήμερα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία υπάρχουν κάποιοι κανόνες για την εργασία, υπάρχουν κανόνες για το περιβάλλον, για την ενέργεια και όταν μιλούμε για μαζική εκβιομηχάνηση θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει ένα υψηλό ε, κόστος της εργασίας στην Ευρώπη, με το οποίο δεν θα πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις. Θα πρέπει να παραμείνουν υψηλοί οι μισθοί και αμοιβέ των εργαζομένων. Ένα τεράστιο θέμα μετά το Brexit είναι ε, τα δημοσιονομικά έσοδα δεν είναι πολλές οι λύσεις, είναι περιορισμένες οι δυνατότητες. Είτε θα έχουμε λιγότερο προϋπολογισμό, επειδή φεύγει το Ηνωμένο Βασίλειο, είτε θα δίνουν περισσότερα οι άλλες χώρες, είτε συνδυασμό των δύο. Ε, ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η γεωμετρία των αντιφάσεων. Ε, άρα πρέπει να υπάρχουν και ήδη πόροι. Όταν γίνεται λόγος για τον προϋπολογισμό, εκεί δείχνουμε και από εκεί κρινόμαστε για το πόσο εμπιστευόμαστε την Ευρώπη γενικά. Μέχρι τώρα τίνουμε να εστιάζουμε ε, στον οικονομικό αντίκτυπο του Brexit. Κατά την άποψή μας έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία να συζητήσουμε για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με την πρόσβασή του στην ενιαία αγορά αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικότερο ως θέμα από το μέγεθος ε, της συνεισφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, της απώλεια και τον τρόπο με τον οποίο θα αναπληρωθεί αυτή. Θα ήθελα να, να πω και σε πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Ε, θα έχουμε ίσως και άλλες ευκαιρίες να συναντηθούμε στο μέλλον ή να απαντήσω και σε άλλες ερωτήσεις σας. Βεβαίως, θα τα ξαναπούμε στη Σόφια, δεν είναι η τελευταία φορά, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων που διοργανώνει η Βουλγαρική Προεδρία και δέχομαι και την πρόσκληση εξ ονόματος της Επιτροπής μας για όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ, για την παρουσίαση και την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε, δεν θα χαθούμε. Πολύ καλή επιτυχία στη Βουλγαρική Προεδρία. Και τώρα συνεχίζουμε το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξή μας, το οποίο είναι μία έκθεση της ομάδας των Πρασίνων, πολιτική συνοχή και κυκλική οικονομία. Η κυκλική οικονομία είναι μία έννοια που έρχεται σε αντίφαση με την παραδοσιακή γραμμική οικονομία. Ε, δηλαδή, το παλιό μοντέλο γραμμικό παραγωγή ήταν κατασκευάζει ένα προϊόν, το χρησιμοποιεί και το πετάς. Ενώ ε, η κυκλική οικονομία σέβεται περισσότερο το περιβάλλον και ε, την σωστή και σόφρονα διαχείριση των φυσικών πόρων. Η πολιτική συνοχή έχει πρωταγωνιστικό ρόλο για να υλοποιηθεί η κυκλική οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις με τον εισηγητή μας, τον κύριο Ντάβορ Σκρλέτς. Θα του δώσω το λόγο. Παρακαλώ τους συναδέλφους που αποχωρούν από την αίθουσα να το πράξουν. Αθορύβως. Έχετε το λόγο, Ευχαριστώ. Θα μιλήσω στα κροατικά. Έχω μία όχι ιδιαίτερα μακροσκελή ομιλία, προκειμένου να αποτελέσει η έναρξη της συζήτησή μας ε, για την έκθεση. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μοιραστώ μαζί σας ε, τις σκέψεις και τις ε, ιδέες που έχω για την κατάρτιση της γνωμοδότησης αυτής. Η κυκλική οικονομία αποτελεί μία από τις ε, πιο σημαντικές δημόσιες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίαση κομισιόν κατά την εντολή της αυτή τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία αποτελούν το κύριο θεμέλιο για την επίτευξη φιλόδοξων στόχων. Επομένως, πιστεύω ότι η έκθεση αυτή έρχεται στη σωστή χρονική στιγμή για να βοηθήσει την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης να αναλύσει τις επιτυχίες της πολιτικής συνοχής κατά την προώθηση της μετάβασης σε ένα νέο οικονομικό μοντέλο κυκλικής οικονομίας. Όμως το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε προτάσεις ε, για την μελλοντική προγραμματική περίοδο. Η κυκλική οικονομία και η πολιτική συνοχής διέπονται από την ίδια λογική, συνεισφέρουν ε, στην ε, προώθηση της οικονομίας των περιφερειών μας. Η Ευρώπη γνωρίζει ότι λείπουν ε, τα, οι ορυκτοί πόροι και ποιοι είναι, ποιος είναι ο αντίκτυπος ε, της χρήσης τους. Φυσικά αντιμετωπίζουν προκλήσεις ε, και οι περιφέρειες και οι τοπικές περιοχές. Στις παραδόσεις μας αλλά και στην καινοτομία μπορούμε να βρούμε λύσεις. Σύμφωνα με την έρευνα και κάποιους υπολογισμούς, το ετήσιο κόστος ε, της ε, γραμμικής οικονομίας κοστίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 7,2 εκατομμύρια ετησίως, δηλαδή 20 φορές τον προπολογισμό πολιτικής ε, συνοχής 2014-2020. Επομένως, πρέπει μέσω της πολιτικής συνοχής να στρέψουμε την Ένωση προς τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Επίσης, πρέπει να αναγνωρίσουμε την ε, σημασία των συνδύων να βελτιστοποιήσουμε την χρήση των υφιστάμενων πόρων ε, και υλικών και να προσπαθήσουμε να σεβαστούμε τους ε, φυσικούς πόρους. Το να άρουμε τις εξωτερικές επιρροές πρέπει να είναι κάτι που θα διέπει το σχεδιασμό των επιχειρηματικών μας σχεδίων θα πρέπει να προωθήσουμε την ε, ψηφιακή τεχνολογία, ε, την ε, επισκευή των προϊόντων, θα πρέπει να αλλάξουμε την εικόνα των πόλεων και των χωριών μας και να καταστήσουμε τις αλλαγές πραγματικές. Η πολιτική συνοχή δεν αφορά μόνο την πολιτική των υποδομών, αλλά ουσιαστικά διαφυλάσσει την κοινωνική συνοχή και την ελληνική στην έκθεση. Εξετάζουμε και την έκθεση της κυκλικής οικονομίας να καταστεί ένας ξεχωριστός στόχος εντός της πολιτικής συνοχής προκειμένου τα νέα επιχειρησιακά προγράμματα να στοχεύουν, να αντικατοπτρίζουν καλύτερα το στόχο αυτό. Επικεντρωνόμαστε και στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ε, που γνωρίζουν την τοπική αγορά και μέσω συνεργασίας με την κοινότητα μπορούν να φέρουν θετικές αλλαγές και να αυξήσουν τη συνειδητοποίηση, την ευαισθητοποίηση για την δυναμική της καινοτομία καθώς και για τις υφιστάμενες βέλτιστες πρακτικές. Θέλουμε να δημιουργήσουμε τοπική αξία, τοπικές θέσεις εργασίας ε, που να είναι ανθεκτικές και να ε, παράγουν προϊόντα που θα μπορούν να ανακυκλωθούν ή να επισκευαστούν. Υπάρχει πολύ μεγάλο δυναμικό που δεν χρησιμοποιείται όπως ε, παραδείγματο χάρη τα βιοδιασπόμενα υλικά που θα μπορούσαν να παραχθούν τοπικά. Αυτό θα μπορούσε να έχει επίπτωση και στην μείωση των λιμάτων. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και πράσινες δημόσιες προμήθειες. Αν ακολουθήσουμε κυκλικές, αρχές κυκλικής οικονομίας στις δημόσιες προμήθειες, μπορούμε ε, να προωθήσουμε αρχές. Ε, επίσης, ε, θα πρέπει να πετύχουμε περισσότερο όφελος για τις ε, τοπικές αρχές. Ε, προβλήματα όπως ε, τα λίμματα στη θάλασσα μπορούν να λυθούν υιοθετώντας και μία μακροπεριφερειακή προσέγγιση γιατί οι μακροπεριφέρειες συχνά αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα με διασυνοριακή δράση. Θα αφιερώσουμε και ένα τμήμα της έκθεσης στη διαχείριση των αποβλήτων θα υιοθετηθεί ε, ουσιαστικά ένα ε, νέο νομοθέτημα που θα αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων. Ο δραστικός διάλογος ε, θα αποτελεί μια πλατφόρμα μέσω των οποίων θα ευαισθητοποιηθούν οι τοπικές κυβερνήσεις σε σχέση με τη σημασία του να ευθυγραμμίσουν με την κυκλική οικονομία project της διαχείρισης των αποβλήτων. Ε, μόνο ένα μικρό μέρος αυτών των σχεδίων χρηματοδοτείται από τα Διευθυντική ταμεία και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Αν δούμε το πώς γίνονται οι επενδύσεις στα κράτη-μέλη, χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες για αλλαγές. Κάποια κράτη-μέλη θέλουν να επενδύσουν σημαντικά ποσά σε ε, διάφορες ε, διάφορα εργοστάσια αποτέφρωσης ε, ή επεξεργασίας ε, λιμάτων, ε, το χάρη σε εργοστάσια που έχουν να κάνουν με την ανακύκλωση. Όμως μια τέτοια προσέγγιση μας μπλοκάρει, μας κρατά μακριά από τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Εδώ καλωσορίζω και τις γνωμοδοτήσεις των Επιτροπών Ήτρε και Ένβη γιατί θα έχουν προσθέμενη αξία για τη δική μας έκθεση σας ευχαριστώ και περιμένω και τα σχόλια των συναδέλφων που θα βελτιώσουν την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους Σκιώδης, ξεκινώντας με τον κύριο Μπόγκοβιτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ τον Ταβόρ για την εισαγωγική του αυτή παρέμβαση και ελπίζω να συνεργαστούμε καλά. Είναι σημαντικό ο τομέα αυτό. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλη πίεση μέρα με την ημέρα σε ό,τι αφορά τους φυσικούς και για πολλούς λόγους. Απλούς. Πρώτα απ' όλα ότι αυξάνουν τον πληθυσμό στον πλανήτη, άρα καταναλώνουν αυτοί οι άνθρωποι περισσότερα τρόφιμα, ενέργεια. Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πιο αποδοτικά και με πιο ευφύ τρόπο η ενέργεια. Και πρέπει να ληφθούν σχετικά μέτρα. Η κυκλική οικονομία ουσιαστικά είναι μια φυσική διαδικασία και χρησιμοποιείται, αξιοποιείται εδώ και πολλά χρόνια γιατί δεν θα βρισκόμαστε εδώ αλλιώ. Υπάρχει πολύ δυναμικό στον τομέα της Γεωργίας για παράδειγμα από το οποίο μπορούμε να αντλήσουμε. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους φυσικούς πόρου. Να μην χρησιμοποιούμε τόσο τα ορυκτά καύσιμα. Και έχουμε πολλέ ευκαιρίε. Όπω αναφέρθηκε Μπορούμε να ακολουθήσουμε καλές γεωργικές πρακτικές. με των καλλιεργιών, για παράδειγμα, η βιοοικονομία επίσης ε, είναι μια άλλη δυνατότητα στον τομέα αυτό. Έχουμε το νόριστο του 2020, έχουμε και κοινοπραξίες. 900 εκατομμύρια ευρώ και άλλα τρία δις από τον ιδιωτικό τομέα για νέα project. Αυτό σημαίνει ότι με την καινοτομία μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη και να παραγάγουμε νέα υλικά, νέες ύλες. Κάτι πολύ σημαντικό είναι να δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας στην Ήπεθρο γιατί γνωρίζουμε ότι η ανάπτυξη της υπαίθρου είναι πολύ σημαντική, <coughs> ιδίως για αυτούς που ζουν εκεί. Με το ορίζοντα 2020 έχουμε τις δυνατότητες να το πετύχουμε. Υπάρχουν όμως και στην κοινωνική πολιτική και στον τομέα της ανάπτυξης της υπαίθρου κονδύλια που μπορούμε να δώσουμε και για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά τη γεωργία, ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι να αλλάξουμε την οτροπία μας και τον τρόπο που λειτουργούμε. Το 1 τρίτο των ε, τροφίμων, για παράδειγμα, τα πετάμε στα σκουπίδια. Νομίζω με αλλαγή των διατητικών μας και τροφικών μας συνήθειών μπορούμε να περιορίσουμε τις πατάλη των φυσικών πόρων ε, και σε τοπικό επίπεδο ε, αυτό που μπορεί να γίνει είναι, παραδείγματος χάρη, η καλύτερη επεξεργασία των αποβλήτων και απορριμμάτων. Αυτό σχετίζεται και με τα ταμεία συνοχής. Έχουν γίνει πολλά και κατά το παρελθόν στον τομέα αυτό. Με τα, ταμεία, με τα κονδύλια συγγνώμη, της συνοχής μπορούν να γίνουν πολλά για τις καλύτερες υποδομές στον τομέα της επεξεργασίας αποβλήτων και απορριμμάτων. Υπάρχουν κονδύλια με τα οποία μπορούμε να βοηθήσουμε τις περιφέρειες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που προβλέπουν διαφορετικά υλικά και διαφορετικές διαφορετικές μέθοδοι παραγωγής. Σε ό,τι διαφορά την ενέργεια. Όχι μόνο σε σχέση με τα χρήση των αποβλήτων, αλλά και σε άλλους τομείς. Στη βιοοικονομία, για παράδειγμα. Έχουμε τη βεθανόλη, βιομάζα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα παράγωγα προϊόντα. Επίσης θέλω να πω ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία να εκπαιδεύσουμε Ιδίω του νέου. Οι νέοι ήδη ε, τα βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα. Από το σχολείο πρέπει να ξεκινήσουμε. Να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψη. Οι τοπικέ κοινωνίε, περιφέρειε έχουν επίση έναν τεράστιο ρόλο να διαδραματίσουν γιατί εκεί γίνονται πολλά στην πράξη. ίσως τα περισσότερα. Στο τοπικό, στο περιφερειακό επίπεδο. Γι' αυτό είναι σημαντικό το Ταμείο Συνοχή, τα διαρθρωτικά ταμεία να συνεισφέρουν ώστε να έχουμε πρόοδο στον τομέα αυτό. Αυτά είχα να πω. Στο μέλλον φαντάζομαι ότι θα μπορέσω να καταθέσω και τροπολογίες για να συνεισφέρω στην πρώτη τη του. Η κυρία Σμόλκοβα, ε, σκιώδη συγγήτρια επίση. ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αν δούμε τι λένε οι στατιστικές για την κυκλική οικονομία, θα καταλάβουμε ότι έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα δεν είναι καλά ούτε για το μέλλον της χλωρίδας και της πανίδας ούτε για την ανθρώπινη υγεία. Θα πρέπει η πολιτική συνοχής και η οικονομία συνοχής να εγγραφεί στην κυκλική οικονομία. Την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια σειρά μέτρων για την κυκλική οικονομία. Ήδη από το 2015 είχαν εξαγγελθεί και εγκριθεί τα μέτρα αυτά. Τώρα αυτό που έχει σημασία είναι να συμφωνήσουν όλα τα κράτη-μέλη για να υλοποιηθούν. Η δική μας πολιτική ομάδα, σοσιαλιστές και δημοκράτες, είχε ένα έγγραφο θέσεων για το πρόγραμμα εργασίας, ε, το οποίο το εκπονήσαμε ήδη από το 2015. Αυτό μου διευκολύνει εμένα τη δουλειά, γιατί ε, μπορώ να σας παρουσιάσω τη θέση της πολιτικής μου ομάδας. Ακούσαμε τον εισηγητή προφορικά. Δεν έχουμε ακόμα κανένα κείμενο στα χέρια μας. Πάντως οι σοσιαλιστές και δημοκράτες θεωρούν ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κονδύλια από τον ορίζοντα 2020 για την οικολογική καινοτομία κυρίως, για την υποστήριξη της έρευνας και της επιστήμης, για περισσότερη ανακύκλωση αλλά και για ε, τη στήριξη των κατασκευαστών ε, ε, για να πληρούν όλες τις προδιαγραφές της ανακύκλωσης. Επίσης, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης να ευαισθητοποιούνται για να κάνουν περισσότερη ανακύκλωση. Έτσι θα αυξηθεί και η απασχόληση. Όταν κάνω λόγο για ανακύκλωση, δεν μιλώ μόνο για το πλαστικό, ας πούμε, ή για το γυαλί ή για τα οικιακά απορρίμματα αλλά αναφέρομαι και στα έπιπλα, για παράδειγμα, στα ρούχα ή και στα διάφορα δομικά υλικά. Εδώ δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τους καταναλωτές. Είναι πολύ σημαντική η στάση των καταναλωτών στην κυκλική οικονομία. Θα πρέπει ο κόσμος να είναι ενημερωμένος, να γνωρίζει περί τίνος πρόκειται, να αρχίζει από το σχολείο ενημερωτική εκστρατεία και με την υποστήριξη μη κυβερνητικών οργανώσεων μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. σε επόμενη φάση να ασκήσουμε πίεση στα κράτη-μέλη έτσι ώστε η κυκλική οικονομία να επιβληθεί. Υπάρχουν καλές πρακτικές και καλά παραδείγματα ήδη από σήμερα. Υπάρχουν κράτη-μέλη όπου κάθε πολίτης παράγει 250 κιλά απορρίμματα το χρόνο. Και είναι ε, απορία άξιου όπω υπάρχουν κρατημέλη που έχουν το τριπλάσιο ανακάτοικο ετησίω. Επίσης δεν θα πρέπει να λησμονούμε τους εργαζομένους στην κυκλική οικονομία, σε αυτούς τους κλάδους. Διότι ακριβώς όσοι ασχολούνται με την επεξεργασία των αποβλήτων έχουν μεγαλύτερους κινδύνους να αντιμετωπίσουν για την υγεία τους. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω την κυρία Τόμασιτς, εξ ονόματος των φιλελευθέρων. Ποιος θα μιλήσει, ο κύριος Βαν Μέλτενμπουργκ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αστροζεβίσιου είναι ο σκιώδη μα, εμεί ανέκαθεν να αναφανδό υπέρ ε, της ε, συνολικής μετάβασης προς μια κυκλική οικονομία. Αυτό είναι σημαντικό για μια μακροπρόθεσμη αηφόρο ευρωπαϊκή ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, αλλά και για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Η Ευρώπη θα πρέπει να σταματήσει να είναι μια κοινωνία ε, των ε, πραγμάτων μιας χρήσεως που πετάμε αδιακρίτως. Θα πρέπει να ανακυκλώνουμε τα πράγματα ε, και να μεταβούμε σιγά σιγά προς την πιο κυκλική οικονομία. Έτσι πιστεύει ο Σκιώδης μας ότι θα ανοίξουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας για περισσότερη απασχόληση και θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Όλα αυτά χρειάζονται θάρρος και πραγματική δράση, αλλά θα πρέπει να είμαστε αρκετά φιλόδοξοι έτσι ώστε να καταλάβουμε ποιε είναι οι προκλήσεις και ποιε οι ευκαιρίες για την κυκλική οικονομία. Βεβαίως την πολιτική συνοχή. Ο σκιώδη ηγητή μα, λοιπόν προσβλέπει και περιμένει την έκθεση αυτή ε, και την ε, γόνιμη συνεργασία και προσωπικά όπως είπα προηγουμένως είναι τεράστιες ευκαιρίες στη λεγόμενη βιοοικονομία. Υπάρχει αυτή η σύμπραξη, το έχουμε ξανασυζητήσει και στην Επιτροπή μας είναι πάρα πολύ ειδικό κλάδος της κυκλικής οικονομίας και θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φαν Πούρχ. Κατάφερε να έρθει σχεδόν στην ώρα της η κυρία Τόμασιτς. Είστε σκιώδης εσείς έτσι, για την κυκλική οικονομία, παρακαλώ. I'm Σας ζητώ συγγνώμη. Έπρεπε να πάω στην Επιτροπή Αλίας. Είχαμε ψηφοφορία. Θα μιλήσω κρατικά. Η σημερινή χρήση των πόρων δεν είναι βιώσιμη. Χρησιμοποιούμε περισσότερες πρώτες ε, ύλες ε, από όσες μπορεί να παράγει ο πλανήτης μας μακροπρόθεσμα. Μέχρι το 2050 κατά μέσο όρο η κατανάλωση θα είναι 6-7 δισεκατομμύρια, κάτι που θα αυξήσει την πίεση στο περιβάλλον. Ο σημερινός τρόπος ζωής μας απαιτεί μεγαλύτερη άνεση, όμως φυσικά αυτό έχει και κάποιο κόστος. Ας δούμε το παράδειγμα των πλαστικών. Σπάνια ανακυκλώνονται. Και απορρίπτοντας το πλαστικό, θέτουμε σε κινδύνο την υγεία των θαλασσών μας. Βλέπουμε τρομερές σκηνές, τόνους απορριμμάτων. Το είδαμε και φέτος. Όμως αυξάνονται οι ποσότητες και είναι ένας όλο ένα και μεγαλύτερος κίνδυνος. Φυσικά αυτό γίνεται όλο ένα και πιο προφανές ε, όταν ε, οι αστικές περιοχές γεμίζουν με απορρίμματα. Αυτό αποτελεί το αποτέλεσμα της χαμηλής διάσπασης ε, του πλαστικού σε μικροσωματίδια. Η κυκλική οικονομία θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο αυτό που προέρχεται από την κυκλική οικονομία που χρησιμοποιεί την αρχή του φτιάχνω, χρησιμοποιώ και πετάω. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τα διπλώματα ευρεσιτεχνία, τους τρόπους ε, Τη ε, χρήση για να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί στην ανακύκλωση. Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία θα πρέπει να συμπεριλάβει την απόκτηση νέα γνώση και να ακολουθούμε και τις νέες εξελίξεις. Ελπίζουμε ότι οι χαράκτες της πολιτικής γνωρίζουν όλα τα δεδομένα και τις εξελίξεις ε, προκειμένου να μπορούν να αναπτύξουν ευέλικτες και κατάλληλες πολιτικές. Θέλω να καλωσορίσω τη δεύτερη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Στην έκθεση αυτή για την κυκλική οικονομία ο οργανισμός κάνει λόγο για μηχανές και νέες τάσεις στην παραγωγή και στη χρήση των πόρων προκειμένου να σεβαστούμε τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Παραδείγματος χάρη έχουμε καινοτομία που σχετίζεται με τα κινητά τηλέφωνα ή με τους εκτυπωτές 3D τους τρισδιάστατους εκτυπωτές. Αυτά μπορούν ε, να ενταχθούν στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία δεν μπορεί να συμβεί χωρίς την υποστήριξη ισχυρών πολιτικών και οικονομικών δομών που θα δίνουν κατευθυντήρες γραμμές για μελλοντικές δράσεις στον τομέα της, της ε, κυκλικής οικονομίας. Η κοινωνία μας αλλά και ο επιχειρηματικό κλάδος θα πρέπει να παρακολουθούν ενεργά τις εξέλιξεις στην τεχνολογία και θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για ανάπτυξη στον τομέα αυτό. Οι κανόνες που διέπουν την κυκλική οικονομία αποτελούν πρόκληση για τα κρατημέλη γιατί θα πρέπει να γίνουν πολλές αλλαγέ. Αυτό δεν θα γίνει ε, χωρίς τις ε, κατάλληλες πολιτικές. Ε, θα πρέπει να τεθούν πρότυπα και στόχοι και φυσικά θα πρέπει να προσπαθήσουμε και να πετύχουμε τους στόχους μας. Θα πρέπει να εισαχθεί και ένα τέλος επιστροφής που θα αποτελέσει κίνητρο. Το ίδιο ισχύει και για την νέα χρήση του ανακυκλώσιμου υλικού. Ε, κυρία Μίχελς, ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Παπαδημούλης χρειάστηκε να φύγει για να πάει σε άλλη επιτροπή να ψηφίσει. Γι' αυτό με χαρά τον αναπληρώ είναι γεγονός. Η πολιτική συνοχής είναι πραγματικά το κλειδί για την επίτευξη της κυκλικής οικονομίας. Παραδείγματα εδώ είναι η ενίσχυση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αποτελεσματική χρήση των πόρων και μια οικονομία με επενδύσεις κλάδους που δεν ε, εκλείουν διοξίδιο του άνθρακα. Για τη δική μας πολιτική ομάδα είναι πολύ σημαντικό στους στόχους να έχουμε μία συνοχή και μία συνεκτικότητα. Πολύ συχνά το συζητάμε και δεν χωράει καμιά αμφιβολία ότι επιδεινώνεται με ταχύς ρυθμούς το περιβάλλον και θα πρέπει αυτό να σταματήσει. Από την άλλη όμως θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όλο και περισσότερο ε, ότι ε, μας ενδιαφέρει να καταργηθούν οι κοινωνικές ανισότητες που είναι και ομολογημένος στόχος της ε, πολιτικής ε, συνοχής. Έτσι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης, θα τονωθεί η επιχειρηματικότητα των νέων και θα έχουμε και πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις στις περιφέρειες. που θα μπορούν να έχουν και πλεονέκτημα από τις ε, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την καλύτερη πρόσβαση σε αυτές. Η κυκλική οικονομία λοιπόν δίνει κατεπληκτικές ευκαιρίες για να τηρήσουμε τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και τη συμφωνία του Παρισιού γιατί οι στρατηγικές κυκλικής οικονομίας μπορεί να συνεισφέρουν ε, προς τα εκεί, τις σχετικές επιπτώσεις στο κλίμα να τις μειώσουν, να τις απαλύνουν γιατί εξ όσων γνωρίζουμε το 67% των εκπομπών αερίων ε, του θερμοκηπίου παγκοσμίω έχουν σχέση με τη διαχείριση ε, υλικών. Αυτό το είπαν και ο εισηγητής και διάφοροι μιλητές. Άρα έχει σημασία σε χώρες που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο να διαδραματίσουν την κυκλική οικονομία, αντίστοιχη πολιτική συνοχή θα πρέπει να έχει επαρκή χρηματοδότηση για την υποστήριξη όλων αυτών των στόχων. Και ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή και τον έφερε. Έχουν πολύ σημαντικό ρόλο εδώ να παίξουν οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις ε, στην ε, ανακύκλωση. Χρειάζονται βελτίωση της βιοοικονομίας, νέα προϊόντα, νέα ε, μορφή θέσεων απασχόλησης, λεγόμενες πράσινες θέσεις εργασίας. Όλα αυτά τα λέει και ο ίδιος ο εισηγητής και τα παρουσίασε και σήμερα εδώ. Έχει σημασία λοιπόν να πούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όλα αυτά δεν είναι κάτι που θα πρέπει να παρασχολούν μόνο τη δική μας Επιτροπή της Περιφερειακής Πολιτικής, αλλά και τη βιομηχανική πολιτική και άλλους κλάδους και άλλες επιμέρους κοινοβουλευτικές επιτροπές. Και θα πρέπει να ενημερώνεται και το κοινό. Για όλα αυτά τέλος να πω ότι η ενίσχυση και η πρόθεση της κυκλικής οικονομίας εγγράφεται θαυμάσια στη στρατηγική κατά του πλαστικού που ε, μας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην περασμένη Ολομέλεια. Αλλά όλα αυτά που συζητάμε και όλοι αυτοί οι στόχοι που θέτουμε για την κυκλική οικονομία και την ανακύκλωση είναι ωραία, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο και δεν είναι το πιο αποτελεσματικό είναι η αποφυγή παραγωγής απορριμμάτων για αποβλήτων. Και εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ίδια έχει κάποια κενά να ανακαλύψει Ευχαριστώ κυρία Νταμάτου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο. Θα συνεργαστούμε πολύ καλά μαζί του, γνωρίζω, σε ό,τι αφορά την οικονομία και σε ό,τι αφορά δηλαδή τον νέο τρόπο να ασκούμε οικονομία. Ξέρουμε ότι το 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τη δεσμή μέτρων για την κυκλική οικονομία για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις, τους ε, καταναλωτές ε, να προβούν σε αυτή τη μετάβαση για μια πιο κυκλική οικονομία, των οποίων οι πόροι θα χρησιμοποιούνται πιο βιώσιμα, αυξάνοντας την ανακύκλωση, την ε, χρήση εκ νέου και να ωφελούν το περιβάλλον. Η πολιτική συνοχής ε, έχει ε, παίξει έναν σημαντικό ρόλο με την κατάλληλη χρηματοδότηση και φαίνεται απαραίτητη χρήση των πόρων αυτών στα διάφορα επιχειρησιακά προγράμματα των κρατών μελών αν ε, και για να ξεκινήσουν και διαπραγματεύσει, για μετά το 2020. Πρέπει να αξιολογήσουμε και τη συνέργεια των κονδυλίων συνοχή ε, με τον ορίζοντα 2020 650 ε, εκατομμύρια ευρώ έχουν εκπονηθεί για διάφορα συγγνώμη, έχουν εκταμιευτεί για διάφορα προγράμματα στη διαχείριση του, μάλλον το έτος 2017, η Κομισιόν παρουσίασε κάποιες νομοθετικές ε, προτάσεις που προέρχονταν από το σχέδιο δράσης και συγκεκριμένα την νομοθετική πρόταση ε, για τα απόβλητα ε, και για τα αγαθά που πολλούνται επιγραμμικά θα ήθελα να σταθώ στην τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων ε, του πακέτου για τα πόβλητα, γιατί χρειάζεται μια σημαντική αλλαγή ε, ρυθμού για να έχουμε αποτελέσματα. Και αυτή η αλλαγή ρυθμού θα πρέπει να γίνει από τα κράτη-μέλη. Πριν ε, ένα μήνα, το Δεκέμβριο του 2017, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε μια συμφωνία για το λεγόμενο πακέτο των αποβλήτων. Σε σχέση με τους στόχους, όμως, η συμβιβασμός δεν είναι αρκετό ε, ε, και είναι ένα βήμα πίσω σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των ε, οικιακών αποβλήτων. Ναι, το νέο ψήφισμα αφορά μόνο τα οικιακά απόβλητα, δηλαδή το 10% αυτών που παράγονται από την βιομηχανική μας οικονομία. Πρόκειται για ένα ντροπαλό βήμα προς τα και εμείς περιμέναμε από το κίνημά μας να γίνει κάτι με περισσότερο θάρρος. Ε, επίσης, σε ό,τι αφορά τις ε, χωματερές, ε, εδώ το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει ανώτατο όριο 5% μέχρι το 2003, ενώ ο τελικός συμβασμός θέτει το στόχο στο 10% και η προθεσμία είναι μέχρι το 2035. Ακυρώθηκαν λοιπόν οι στόχοι που είχαν προτεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, εκ νέου χρήση των προϊόντων που στόχευαν στο να δημιουργηθούν νέε θέσει εργασία και να μειωθούν τα απόβλητα. Επίση, κάτι άλλο που αφορά τα απόβλητα των τροφίμων. Σήμερα με την Κομισιόν ε, κάθε χρόνο σε όλα τα κράτη πετιούνται 88 εκατομμύρια τόνοι ε, τροφίμων και ε, υπολογίζεται ότι αξίζει όλα αυτά 143 δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, μόνο ε, παρόλα αυτά δέχτηκε το Συμβούλιο να μειώσει κατά 30% μέχρι το 2015 αυτά τα απόβλητα και μέχρι το 2030 5% παραπάνω. Όμως δεν είναι δεσμευτική αυτή η στόχη και τα κράτη-μέλη απλώς θα πρέπει να στείλουν μια έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό απλώ αποτελεί ένα παράδειγμα που δείχνει πω η πολιτική βούληση θα πρέπει να είναι πολύ πιο φιλόδοξη σε όλα τα επίπεδα με πραγματικό πρωταγωνισμό και εμπλοκή τη τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αγωνιστούμε για πιο φιλόδοξου στόχου για να δημιουργήσουμε νέε θέσει εργασίε και να ε, μειώσουμε τόνου διοξιδίου, διοξιδίου του άνθρακα εμείς ε, το οφείλουμε και στους εαυτού μας αλλά και στις μελλοντικέ γενιές. Ε, πώς ε, λοιπόν θα διορθώσουμε αυτό το συμβιβασμό σε ό,τι μας αφορά φυσικά, σε ό,τι αφορά τη δική μας επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτή την έκθεση, να κάνουμε κάποιες προτάσεις για μετά το 2020 θα μπορέσουμε να θέσουμε περισσότερους πόρου στο συγκεκριμένο στόχο, παραδείγματος χάρη να έχουμε περισσότερους πόρους στην περίπτωση περίπτωση της κατάργησης ε, των χώρων υγειονομικής ταφής. Ε, θα είναι κάποιες προτάσεις αυτές που θα κάνω κατά τη συνάντηση των σκιωδών. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ακόμη ονόματα έχω. κύριος ε, Ροπέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι πάρα πολύ που συμφωνούμε γενικά σε αυτό το θέμα. Έχει έρθει η ώρα να ε, επιδιώξουμε περισσότερα, με μεγαλύτερη φιλοδοξία. Ελπίζω να αποδώσει αυτή η προσπάθεια έχουμε αναλάβει την υποχρέωση στην Ευρώπη να εγκαταλείψουμε ε, τα ορυκτά καύσιμα. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε λοιπόν και για τις ημερομηνίες τώρα και για τη μετάβαση ε, σε μια κυκλική οικονομία. Διάβασα κάπου μια είδηση και χάρηκα πολύ ε, που έλεγε ότι οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι από τις αρχές του έτους ε, λειτουργούν με πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Δηλαδή 100% το ηλεκτρικό ρεύμα, ε, όχι στη Γερμανία, συγγνώμη, στη Λιθουανία, ε, τα τρένα κυκλοφορούν με ρεύμα που έχει παραχθεί με οικολογικό τρόπο. Ορίστε, γιατί να μην είναι αυτό ένα παράδειγμα προς μίμηση στα άλλα κράτη-μέλη και να υποχρεούνται οι σιδηρόδρομοι να ε, το ακολουθήσουν αυτό. Ή ας πούμε ε, οι δρόμοι να φωτίζονται ε, στους δήμους και της κοινότητας, ο δημόσιος φωτισμός δηλαδή, από ηλεκτρικό ρεύμα που έχει παραχθεί με οικολογικό τρόπο, το λεγόμενο πράσινο ρεύμα. Είναι καλές αυτές οι πρωτοβουλίες. Και θα πρέπει να υποχρεούνται και οι εταιρείε ηλεκτρικής ενέργειας να αγοράζουν ε, αυτό το ρεύμα που παράγουν ε, με οικολογικό τρόπο ε, όσοι έχουν φωτοβολταϊκά ας πούμε ή τέτοια μορφή παραγωγής και όχι κατά ανάγκη ακριβότερα. Ευχαριστώ κύριος Φανίστερ Ρόι. Χαίρομαι πάρα πολύ, Πρόεδρε, με αυτά που ακούω. Πολύ μεγάλη συναντήληψη και υποστήριξη αυτής της προσέγγισης και εγώ θα ήθελα να ζητήσω ε, με την άλλη έκθεση να τα δούμε και αυτά ε, την έκθεση που θα ψηφίσουμε το Φεβρουάριο το Μάρτιο για την ε, ε, πολιτικής συνοχής να συνάδει με τη Συμφωνία για το Κλίμα του COP21. Να είναι ένα συνολικό πακέτο, πούμε, μια δέσμη. Και να ακολουθεί ε, τη Συμφωνία του Παρισιού που να φτάνει ε, σε κάθε γωνιά της Ευρώπης, σε όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις. Πολύ καλή η έκθεση αυτή και είχαμε και την έκθεση σοσιαλιστών και δημοκρατών. Εγώ είμαι περήφανος για ε, τις προσπάθειες αυτές. Ακούσαμε ε, τα ποσά ε, ε, που καταβάλλονται στις χώρες της συνοχής για την ανακύκλωση για την κυκλική οικονομία. Υπάρχουν χώρες όμως που η ανακύκλωση δεν φτάνει το 10%, δεν 90% των ε, αποβλήτων καταλήγουν στις Εδώ είναι ένα πράσινο κεφάλαιο και χωρίς να επιβαρύνονται οι πολίτες και οι καταναλωτές μπορούμε να κάνουμε τεράστια βήματα. Υπάρχουν οι τεχνολογίες. Ας είμαστε λοιπόν αισιόδοξοι και μια τελευταία παρατήρηση. Κάτι που μου κάνει εντύπωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα έκανε μια πρόταση για τον κανονισμό για τα πλαστικά. Οι πολίτες δεν τα γνωρίζουν αυτά τα προϊόντα. Υπάρχουν ε, βιοδιασπόμενα υλικά και πλαστικά ε, τα οποία είναι νέα υλικά ας πούμε αλλά ο κόσμος δεν τα γνωρίζει όταν έχεις το παιδί σου και παίζει στην παραλία ε, με ένα τέτοιο κουβαδάκι άμα του πέσει στη θάλασσα μετά από 9 μήνες ξέρω εγώ έχει αποδομηθεί και δεν είναι πλαστικό που ρηπαίνει τους ωκεανούς αλλά οι πολίτες δεν τα ξέρουν αυτό ότι υπάρχουν νέα υλικά, νέες δυνατότητες χρειάζεται επικοινωνία, ενημέρωση, διαφήμιση για να ενισχυθεί και ο πολίτης και να αγοράζει με τα λόγου Ευχαριστώ πολύ. Α, ο κύριος Φανής ήταν ο τελευταίος ε, από τους βουλευτές μέλη της Επιτροπής μας. Ε, θα ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, κ. Μιλοντίνοβα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πραγματικά είναι πολύ θετικά αυτά που άκουσα. Οι απόψεις για την κυκλική οικονομία και για το πόσο σημαντική είναι για μια βιώσιμη μετάβαση. Είναι απόψη με βρίσκουν σύμφωνοι. Εμείς ε, ε, θεωρούμε ότι η πολιτική συνοχή ε, κάνει ήδη πολλά για την ε, κυκλική οικονομία. Είμαστε υπέρ του πακέτου. Όταν προτάθηκε αυτό το πακέτο ήδη βέβαια είχαν κυκλοφορήσει δικοί μας κανονισμοί, αλλά έχουμε τη διαχείριση των αποβλήτων, την ερική χρήση των πόρων, έρευνα καινοτομία, τη στήριξη των επιχειρήσεων, να έχουν δηλαδή όλα αυτά. Τη διαχείριση των αποβλήτων ε, για δεκαετίες την υποστηρίζουμε μέσω της πολιτικής συνοχής. Άρα πολλά έχουν γίνει. Φυσικά και υπάρχει πολύ μεγαλύτερο δυναμικό και πολλές δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης και ανάπτυξης. Θα ήθελα να εστέσω σε δύο πτυχές. Η πρώτη πτυχή είναι επενδύσεις στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Πάνω από 5 δις ακούσαμε ότι είναι το ποσό. Αυτό είναι πολύ θετικό. κάτι ανάλογο με την περίοδο προγραμματισμού την προηγούμενη. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι υπάρχει αλλαγή προς την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση. Δεν μιλάμε δηλαδή για τις ηλικές υποδομές μόνο, αλλά και για μηχανισμούς συλλογής διαλογής, αποκομιδής, ανακύκλωσης. Δηλαδή πιο πολύ στο πώς ε, θα βοηθηθεί ο κόσμος επιτόπου αυτήν την εστίαση σε ό,τι αφορά τη διάθεση των αποβλήτων. Υπάρχουν ακόμη ανάγκες σε υποδομές και μεγαλύτερες μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, ιδίως για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Αναφέρθηκε το ζήτημα των χωματερών. Για τη νέα αυτή περίοδο προγραμματισμού έχουμε την εκ των προτέρων αιρεσιμότητα που σχετίζεται με τα σχέδια διαχείριση αποβλήτων. Οι προκλήσει είναι μεγάλε βέβαια, γιατί φυσικά και τα κράτη-μέλη ήθελαν να έχουν αυτά τα σχέδια και έπρεπε να έχουν αυτά τα σχέδια διαχείριση αποβλήτων. Ο λόγο που διασυνδέουμε αυτά τα δύο είναι είναι να έχουμε περισσότερη ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση Έχουμε την πυραμίδα να πούμε για τις χωματρές. δεν έχω δει κάτι. Νομίζω ότι είναι θετικό που υπάρχει αυτή η ευθυγράμμιση των επενδύσεων. Με το κεκτημένο το ενωσιακό και σε αυτό το θέμα. Έχουμε επίσης μεγαλύτερη υποστήριξη στη διασυνορική και μακροπεριφερειακή συνεργασία. κυκλική οικονομία είναι παρούσα στις δράσεις μας. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι η υποστήριξη που παρέχουμε και στην καινοτομία. Έχετε ακούσει και ξανακούσει την ε, ευφύ εξειδίκευση. Η διαδικασία από κάτω προς τα πάνω. 41 δις είναι το κατά που για αυτό το θεματικό στόχο. Γνωρίζουμε ότι η κυκλική οικονομία επιλέγει από τις περιφέρειες όπως και η ενεργειακή, μάλλον όπως και η αποδοτική διαχείριση, η βιωσιμότητα των πόρων. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα ε, ε που προέρχεται από τις ίδιες περιφέρειες. Η βιοοικονομία ήταν άλλο θέμα που αναφέρθηκε και που εντάσσεται στην εξειδίκευση. Η Ευρώπη έχει λοιπόν αυτή την ευκαιρία. Ξέρουμε ότι η Κίνα δεν φαίνεται να θέλει να εισαγάγει πλέον απόβλητα από την Ευρώπη, πλαστικά απόβλητα. Πρέπει λοιπόν να κατασταθεί το πλαστικό με άλλα προϊόντα, τα βιοπροϊόντα, τα βιοπροϊόντα της βιοοικονομίας. Αυτή είναι μια πτυχή της εφίους εξειδίκευσης. επιπλέον τη παραδοσιακή υποστηρίξη υποδομέων, στις Ήδη λοιπόν έχουμε κάνει μια σημαντική συνεισφορά όπως πρέπει και τώρα θα πρέπει να δούμε όλα αυτά πώς θα οδηγήσουν σε μια πραγματική μετάβαση της οικονομίας μας. Σε όλη τη διάρκεια αυτής της περίοδου προγραμματισμού. Αλλά ίσως και σε μελλοντικές περίοδους. Η κυκλική οικονομία πάντω είναι άκρο σημαντική για τι πολιτικέ μα και για τι περιφέρειε συνολικά. Γι' αυτό είναι και σημαντική άλλωστε για τι πολιτικέ μα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σκάρλετ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. θέλω να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου. για τις ε, σημερινές τους ε, παρεμβάσεις. Και σε αυτή την χρονική στιγμή αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι σαφές ότι πρέπει να γίνει μια ξεκάθαρη διασύνδεση της πολιτικής συνοχής με την κυκλική οικονομία. Και η δημογραφική πολιτική όμως πρέπει να ληφθεί υπόψη. Διότι πολλές χώρες που είναι δικαιούχοι των κονδυλίων συνοχής έχουν το πρόβλημα το ότι οι ναι, νέοι εγκαταλείπουν την Ήπεθρο ή ακόμη και τις πόλεις γιατί πηγαίνουν στο εξωτερικό, επειδή δεν μπορούν να βρουν ντόπιε θέσει. Και εκεί μπορεί να παρέμβει η κυκλική οικονομία. Ακούσαμε την άποψη της ε, Κομισιόν. Μίλησε για την ειδική εξειδίκευση και ότι αυτό είναι σημαντικό να περιληφθεί η στρατηγική της αφιούς εξειδίκευσης. Είναι ένα από τα εργαλεία που πρέπει να έχουμε υπόψη. Έτσι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την οικολογική περιβαλλοντική καινοτομία και την ε, ανάπτυξη νέων υλικών που θα μπορούν να κυκλούνται εύκολα. Επίσης θα παραγάγουμε πιο ε, καλά νέα προϊόντα που θα μπορούν να επισκευάζονται, θα είναι πιο βιώσιμα. Η κυκλική οικονομία πρέπει να ενταχθεί και στο τομέα των δημοσίων προμηθειών. Έτσι ο δημόσιος τομέας και το τοπικό επίπεδο θα αποτελέσουν κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης. Ο διωτικός δε τομέας θα μπορέσει να λάβει πρωτοβουλίες επίσης. Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης πρόσφατα ενέκρινε ένα πρότυπο για τις βιώσιμες επιχειρήσεις. ISO 9001 και, άλλες, και άλλα πρότυπα περιβαλλοντικά αλλά εδώ έχουμε και άλλα πρότυπα που έχουν να κάνουν τον ιδιωτικό τομέα. Οι αρχές της κυκλικής οικονομίας είναι παρούσες και στα δύο αυτά είδη προτύπων. Ευχαριστώ πολύ και θα συνεργαστώ ευχαριστώ με τους ε, σκέφτες στο Μάρτιο θα παρουσιάσετε, αν κατάλαβα καλά, το σχέδιο εκθεσή σα. Μάλιστα. Οπότε θα ψηφίσουμε κατά ψηφιδότητα το Μάιο. Καλή επιτυχία λοιπόν και καλή δουλειά και περνάμε στο επόμενο σημείο της μερικής διάταξης. Πρόκειται για τη γνωμοδότηση για την απαλλαγή για το 2016, Γενικός προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού Επιτροπικών το προετοιμάζει την έκθεσή τη για τη χορήγηση απαλλαγή στην Κομισιόν για την εφαρμογή του προπολογισμού 2016. Η Ρέτζη καταρτίζει μια γνωμοδότηση και εισηγητρία είμαι εγώ. Σήμερα θα παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδοτησή μου που επικεντρώνεται κυρίω στη μείωση του εκτιμόμενου επίπεδου λάθο ε, στον τομέα των δαπανών και στις κυρίες πηγές των επομενών λαθών στις προκλήσεις που έχουμε για την δημοσιονομική εφαρμογή στην σημερινή προγραμματική περίοδο. Θα πρέπει να ψηφίσουμε την νομοδοτησή μας το Φεβρουάριο στη Ρέτζη. Γι' αυτό θα παρουσιάσω σήμερα το σχέδιο γνωμοδότησης και αναμένουμε τις τροπολογίες μέχρι τις 12 το μεσημέρι στις 30 Ιανουαρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Και τώρα θα μιλήσω βουλγαρικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω την ευχαρίστηση να σας παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότησης της Επιτροπής μας για την απαλλαγή του προπολογισμό τη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρετε ότι αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα τη πολιτική ε, συνοχή μετά την ετήσια έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Θα ήθελα να παρουσιάσω και εγώ την γνωμοδότηση ως ε, εισηγήτρια. Σημειώνω ότι όπως βλέπουμε έχουμε μία μείωση του ποσοστού λάθους από 5,2 το 2015 σε 4,8 το 2016. Αυτό δείχνει μία συνολική βελτίωση των διορθωτικών δράσεων των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για πρώτη φορά, μάλιστα, τα τελευταία χρόνια, το ελεγκτικό συνέδριο γνωμοδοτεί με επιφύλαξη σε σχέση με την νομιμότητα και την ορθότητα ε, των πράξεων που αφορούν τον προπολογισμό του 2016. Όμως η έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου μας δείχνει ότι τα κράτη-μέλη είχαν αρκετό χρόνο και ευκαιρίες να διορθώσουν λάθη πριν την επιβολή των διορθώσεων. Επομένως, το ποσοστό λάθους θα μπορούσε να είναι πολύ χαμηλότερο από το όριο σημαντικότητας. Επομένως, θα μπορούσε να έχει γίνει προσπάθεια για να αποφεύγεται το υψηλό ποσοστό λαθών. Πολλά από τα λάθη έχουν να κάνουν με τις κρατικές ενισχύσεις. Καλούμε λοιπόν την Κομισιόν να αναλάβει προληπτική δράση για να εφαρμοστούν οι σχετικοί κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Ανησυχούμε για το ότι μόνο το 77% των ε, αρχών, των αρμοδίων αρχών για την εκτέλεση των προγραμμάτων έχουν διοριστεί από τα κράτη-μέλη. Καλούμε λοιπόν τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν να συνεργαστούν για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Η γνωμοδότηση εκφράζει την ανησυχία της σε ό,τι αφορά την ε, καθυστέρηση της εφαρμογής ε, των προγραμμάτων. Το 2016 το συνολικό ποσό των δημοσιονομικών δεσμεύσεων έφτασαν τα 238 δισεκατομμύρια ευρώ λόγω των καθυστερήσεων αυτών. Αυτές οι αδυναμίες ε, θα πρέπει να ξεπεραστούν κατά το σχεδιασμό του επόμενου πολιτικού δημοσιονομικού πλασίου. Λαμβάνουμε υπόψη τη στρατηγική έκθεση 2017 για την ε, εφαρμογή των ε, Ευρωπαϊκών Διευθυντικών και Επενδυτικών Ταμείων. Οι πόροι των ταμείων αυτών φτάνουν τα 278 δισεκατομμύρια ευρώ. Με άλλα λόγια, η εφαρμογή έχει καλύψει τους στόχους της ε, και φαίνεται η πρόσθετη αξία για όλες τις περιφερειές, τις περιφερειές της Ευρώπης. Μόνο 75% ήταν ε, το μέσο ο μέσος συντελεστής εκταμίευσης, το μέσο ποσοστό εκταμίευσης για τα ε, χρηματοδοτικά μέσα στα τέλη του 2015. Πιστεύουμε ότι μια αναθεώρηση του χρηματοοικονομικού μηχανισμού θα βελτιώσει, θα συνεισφέρει συγγνώμη την απλούστευση και τη βελτίωση των, της χρήσης των κονδυλίων κατά τη σημερινή προγραμματική περίοδο. Επίσης, απευθύνουμε έκκληση στην Κομισιόν να αναθεωρήσει την αποτελεσματικότητα των δικτών που χρησιμοποιούνται και καλούμε την Κομισιόν να βελτιώσει το συνολικό σύστημα μέτρησης της εφαρμογής και των επιδόσεων για την περίοδο μετά το 2020. Αυτό ήταν το κείμενο της ε, γνωμοδότησής μου που σας ανέγνωσα και θα δώσω τώρα το λόγο στους και οδησίγητες Εξ του κυρίου Ντόιτς, ε, Βέλη, θα μιλήσω ουγγρικά εγώ. Ε, θα ήθελα λοιπόν, ε, εξ του σκιώδη συγητού μας, να σας αναφέρω μερικά πράγματα. Δυστυχώ ο κύριο Ντόιτ κολλείται και δεν μπορεί να παρευρεθεί σήμερα. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο και θετικό ε, ότι χρόνο με το χρόνο μειώνεται το σφάλμα. Ε, καλύτερο θα ήταν να μειωθούν και τα διάφορα διοικητικά εμπόδια και το διοικητικό άχθος και εκεί να δείτε πόσο θα μειωθεί το ποσοστό σφάλματος. Θα ήθελα να θυμίσω ότι το γεγονό ότι κάποιος δεν ανταποκρίνεται στους κανόνες και υπάρχει κάποια παρατυπία, αυτό δεν σημαίνει ατασταλία αυτόματα και απάτη. Έτσι, όταν κάποιος δεν συμμορφώνεται προς του κανόνες, δεν σημαίνει ότι υπάρχει δόλος και πρόθεση. Ε, άρα θα πρέπει να είναι έσχατη λύση η επιβολή κυρώσεων τύπου αναστολή πληρωμών. Επίσης ήθελα να πω ότι τα κράτη-μέλη παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, πρωταγωνιστικό θα έλεγα, στις επενδύσεις και στην ε, ανάπτυξη των δυνατοτήτων για τι ε, επενδύσεις αυτές. Θα πρέπει να ανταλλάσσουμε βέλτιστες πρακτικές. Σε ό,τι αφορά ε, τη βελτιστοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων, συμφωνώ απολύτω με τη συντάκτρια τη γνωμοδότησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά στην περιφερειακή ανάπτυξη ε, είναι πολύ μεγάλη σημασία των επιδοτήσεων, δηλαδή των ε, κονδυλίων που διατίθεται χωρίς να πρέπει να επιστρέφονται. Γιατί κάθε επένδυση δεν ε, αποφέρει και κέρδος ή ακόμα και όταν είναι κερδοφόρα αυτό δεν μπορεί πάντα να υπολογίζεται εκ των προτέρων. Αυτά θα κάνουμε τροπολογίες, συμφωνούμε γενικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βόν είναι ο επόμενος ε, σκιώδης, τον οποίο και δεν βλέπω, η κυρία Τόμασιτς. Τι άλλο να προσθέσω εγώ, δεν έχω πολλά πράγματα να πω. Εσείς τα είπατε όλα. Είναι θετικές οι εξελίξεις, τα μέτρα απέδωσαν. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε. Η κυρία Μίχελς. Μπορώ και εγώ να συμφωνήσω, κυρία εισηγήτρια. Το σχέδιο γνωμοδότησή σας ε, περιλαμβάνει τα σημαντικότερα σημεία, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα. Ε, δεν ε, εκταμιεύονται με ικανοποιητικό τρόπο τα κονδύλια. Το 2017 επιστράφηκαν κονδύλια ε, αναπορόφητα στα κράτη-μέλη. Το συζητήσαμε και εδώ αυτό και ελπίζουμε την αλλαγή ε, του δημοσιονομικού κανονισμού να μειωθεί ακόμα περισσότερο το ποσοστό σφάλματος αλλά να αυξηθεί και από ροφητικότητα. Θα ήταν όμως λάθος να ε, συμπεράνει κανείς από τη χαμηλή απορροφητικότητα ότι δεν υπάρχουν ανάγκες. Άρα δεν τα απορροφούν τα κονδύλια. Υπάρχουν τεράστιες ανάγκες οικονομικές και κοινωνικές και είναι πολυτέλεια να τα χάνουμε. Ακριβώς σε χώρες ε, που είναι λιγότερο ανεπτυγμένε. Και είναι υψηλό το ποσοστό των κοινοτικών ε, κονδυλίων ε, σε σχέση με τη συνολική περικοδότηση. Και έχει τεράστιες συνέπειες το ε, να μην γίνονται αυτές οι επενδύσεις γιατί δεν μπορούν να προχωρήσουν τα έργα που έχουν προγραμματιστεί. Νομίζω ότι είμαστε σε σωστό δρόμο και ελπίζω να καταλήξουμε σε μια καλή απόφαση για την απαλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο uh, Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Είναι ισορροπημένη οι γνωμοδότηση αναφέρονται τα σημαντικότερα θέματα. Θα πρέπει να επαγρυπνούμε στο να συνεχίσουμε την καταπολέμηση της απάτης και να είμαστε φιλόδοξοι στο να μειωθούν περαιτέρω το ποσοστό, το λάθος να ανοιχνεύουμε τις απάτες και τις παρατυπίες. Θα πρέπει να ε, ενδυναμώσουμε και τη συνεργασία μας με την Transparency International. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νταμάτου. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με πολλά από τα σημεία που εξέφρασε η Πρόεδρος και συγκεκριμένα ε, το ποσοστό λάθους ε, που υπογραμμίζεται από το Ελεκτικό Συνέδριο στην έκθεση του 2016. Πολύ καλό το υπήρχε μείωση, όμως ε, το 5,2 του 2015 στο 4,8 του 2016. Παρ' όλα αυτά πρέπει να διαπιστώσουμε ότι και πάλι είμαστε πάνω από το αποδεκτό του 2% που είναι το σχετικό κατόφλι. Να θυμόμαστε ότι μιλάμε για χαμηλά ποσοστά, αλλά μιλάμε για μεγάλα ποσά και συνοχή παραμένει ο τομέας όπου έχουμε το υψηλότερο ποσοστό λάθος. Μπορούμε και να τα κάνουμε καλύτερα και πρέπει η Κομισιόν σε μία από τις απαντήσεις της υπογραμμίζει ότι τα project που χρησιμοποιούν τα απλοποιημένες ε, συναλλαγέ υπόκειται σε λιγότερα λάθη. Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια η Κομισιόν έχει προωθήσει την χρήση στο πλήσιο τη πολιτική συνοχή και τη αγροτική ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν εμεί συμφωνούμε με κάτι τέτοιο. Φαίνεται ότι αποδεικνύεται στο πρώτο αυτό στάδιο ότι αυτέ οι απλουστευμένε, με τι απλουστευμένε επιλογέ, οι δικαιούχοι και οι οργανισμοί πληρωμών μπορούν να μειώσουν το διοικητικό άχθο και να επικεντρωθούν περισσότερο στα αποτελέσματα συγκεκριμένα όταν τέτοιες επιλογές ε, βασίζονται ε, στο ότι βλέπουμε ε, πραγματικά αποτελέσματα από τα έργα. Όμως ε, υπάρχουν ε, ανησυχίες ε, στο ρυθμό, στον πολύ αργό ρυθμό υλοποίησης του σημερινού προγραμματισμού. Έχουμε και τον κανόνα νη συν 3, βάσει του οποίου δόθηκαν σημαντικά ποσά στα διάφορα κράτη-μέλη. Στον προγραμματισμό μετά το 2020, ο κανόνας νη συν 2 πάλι θα καταργηθεί έτσι λοιπόν ε, δεν ε, θα μπορούν να εγκρίνουν επιχειρησιακά προγράμματα τα κράτη-μέλη και να διορθώσουν τα λάθη. Ξέρουμε ήδη αυτό τι σημαίνει και έχουμε δει τα ζωφερά αποτελέσματα του, της προγραμματικής περίοδου 2007-2013 ότι υπήρχε νέος ε, προγραμματισμός και μεγάλες δαπάνες καθυστερημένη οθέτηση του κανονισμού έπαιξε μεγάλο ρόλο στη συσσόρευση των καθυστερήσεων ε, γιατί το να λανθάνει κανείς είναι ανθρώπινο αλλά το να μένει στα λάθη του είναι διαβολικό. Ε, ε, και για να κλείσω ε, το ελεκτικό συνέδριο μας λέει ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2015 είχε χρησιμοποιηθεί μόνο το 70% ε, των ε, χρηματοδοτήσεων μέσω των ταμείων ΕΤΠΑ και ΕΧΤΑ. Το ελεκτικό συνέδριο μας λέει ότι πολλά κράτη-μέλη ακόμη και ε, αν παραταθεί η περίοδος ε, δεν θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν πλήρως τις πρικοδοτήσεις. Ε, ένα ποσοστό εκταμίευσης κάτω του 100% σημαίνει ότι δεν εκμεταλλευόμαστε πλήρως αυτά τα εργαλεία η Κομισιόν απάντησε ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση στον νέο προγραμματικό κύκλο με τη μεγαλύτερη εμπειρία των ε, αρχών διαχείρισης. Όμως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για την περίοδο μετά το 2020. Ευχαριστώ. Κύριε Βόν, είστε έτοιμος να πάρετε το λόγο. Yeah, thanks, Sorry, I was a... Uh, Συγγνώμη που καθυστέρησα. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω για την έκθεση που δείχνει ότι το ποσοστό σφάλματος έχει μειωθεί κατά τη, όπως και για την πολιτική συνοχή. Αυτή είναι η τάση, πτωτική. Ίσως όμως ε, να είναι αρκετά αισιόδοξε οι προβλέψει. Το λέω ω πρώτο αντιπρόεδρο τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, η οποία υποστηρίζει ότι εστιάζουμε πολύ στα ζητήματα συμμόρφωσης, αν έχουν ε, μπει και τσεκαριστεί τα τετραγωνίδια κτλ. Αν δεν έχουν, ε, βάζουμε λάθος. Θα πρέπει να δούμε ε, περισσότερο τις επιδόσεις, ε, να μετράμε αυτό στο μέλλον και τα κονδύλια τα οποία δίνονται για project διάφορα και έργα να αποδίδουν. Και αυτό με φέρνει στο δεύτερο σχόλιο που ήθελα να κάνω, ότι στο μέλλον όταν ε, θα εξετάσουμε τους κανόνες για το επόμενο πολιέτης ε, δημοσιονομικό πλαίσιο και τον προσεχή κανονισμό συνοχής, ε, νομίζω ότι για εμάς θα είναι σημαντικό ναι με να μειωθεί το ποσοστό σφάλματος, αλλά να εστιάσουμε περισσότερο στην επίδοση, την απόδοση ώστε πραγματικά να δίνει αποτελέσματα η πολιτικής συνοχής. Επίσης, ε, σε ό,τι αφορά την απλούστευση των κανόνων, αυτά τα λέμε συνεχώς στην Επιτροπή μας. θα πρέπει να είναι μια ενιαία δέσμη ε, κανόνων, απλουστευμένες επιλογές κόστου, το e-cohesion κτλ. Καλό είναι να υπάρχει απλούστευση. Αυτό είναι πολύ καλό για τις δικαιούχους, για τις αρχές των χωρών, αλλά και για τον προϋπολογισμό της Ένωσης και φυσικά για το ποσοστό σφάλματος. Όλα αυτά είναι τα ζητήματα που θα πρέπει να μας απασχολούσουν και πρέπει να σας πω ότι με ικανοποιεί έκθεση γιατί εστιάζει και στο ποσοστό σφάλματος, αλλά δείχνει και προς το μέλλον σε σχέση με κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν. Ευχαριστώ πολύ. πρόεδρε. υπάρχουν άλλα σχόλια. Όχι, θα δώσω τότε το λόγο στον εκπρόσωπο τη ευρωπαϊκή Επιτροπής. Είναι η κυρία Κλοντίν Γκερή. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Let me thank you for your, uh, quite Είναι ισορροπημένη η πρόταση γνωμοδότηση για την πολιτική συνοχή επισημαίνει και τονίζει τις βελτιώσεις που είχαμε σε ό,τι αφορά τα ποσοστά σφάλματος τα τελευταία τρία χρόνια. Το ποσοστό σφάλματος πλέον έπεσε κάτω του 5% και αυτό για πρώτη φορά για την περίοδο 7-13 και θα πρέπει να πούμε ότι και οι διαρθωτικές δράσεις της Κομισιόν των Κατών μελών απέδωσαν τα δέοντα. Θέλω να προσθέσω ότι οι νέες απαιτήσει για την περίοδο 14-20 θα πρέπει να οδηγήσουν και σε περαιτέρω μείωση του ποσοστού σφάλματος. Επειδή έχουμε τους πιστοποιημένους αιτήσους λογαριασμούς και την υποχρέωση, το πολυματικό ποσοστό σφάλματος να είναι κάτω από το 2% κατοφλίου materiality threshold. Αυτό είναι ε, σημαντικό σε σχέση με τον πολιτικό χαρακτήρα που είχαν οι προηγούμενες περίοδοι προγραμματισμού. Ήδη βλέπουμε τα αποτελέσματα των νέων αυτών απαιτήσεων στους πρώτους λογαριασμούς που πήραμε πέρυσι το Φεβρουάριο. Τα ποσοστά σφάλματος που αναφέρθηκαν πραγματικά ήταν πολύ χαμηλότερα από το 2%. Τώρα θα ήθελα να υπογραμμίσω ορισμένα στοιχεία προς ε, εσάς, προς ενημέρωσή σας. Θέλω να στήσω μια αλλαγή στο σημείο 3 που μιλάει για τις κρατικές ενισχύσεις. Και πώς επηρέασε τα πράγματα το ποσοστό σφάλματος εκεί. Δεν είναι αληθές όπως το γράφετε ακριβώ, γιατί πράγματι αναφέρθηκε από το ελληνικό συνεδρίο ότι υπάρχουν κάποια σφάλματα σε σχέση με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Δεν ποσοτικοποιήθηκαν όμω τα σφάλματα, που σημαίνει ότι δεν επηρεάζουν οι κρατικέ ενισχύσει. το ποσοστό σφάλματο για φέτο. Το επιλέξιμο κόστος είναι το κριτήριο και οι δημόσιε συμβάσεις και έπειτα οι δικαιούχοι και οι επιλέξιμοι φορεί. Αυτό είναι μια σημαντική αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Όπου κρατικές ενισχύσεις και δημόσιες ε, Προμήθεια για παράδειγμα το 2014 ήταν η βασική πηγή σφάλματος. Ζητείτε α, προληπτική δράση για την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων από την Κομισιόν και εγώ θα σας παραπέμψω στο σχέδιο δράσης ε, της Κομισιόν που επικαιροποιήθηκε πρόσφατα. Πέρυσι το παρουσίασε στην ΚΟΝΤ και ο γενικός μας ε, διευθυντής σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις ε, στην εφαρμογή των ε, ισχυών προγραμμάτων που τρέχουν για τους ορισμούς. Θα ήθελα να πω ότι σε ό,τι αφορά το designation του ορισμούς έχουμε ένα ποσοστό 87% που καλύπτει το 98% των εδρών, των τοποθεσιών. Δεν είναι δηλαδή θέμα πλέον οι ορισμοί. είχαμε ένα ποσοστό επιλογής 44%. Ε, Επιτόπου. Και αυτό θα μεταφραστεί σε αιτήσεις πληρωμών σύντομα. Σε ό,τι αφορά τα μέσα χρηματοδότησης. 75% αναφέρει το συνεδ... όταν συνέταξε την εκθεσή του. Το ποσοστό αυτό πλέον είναι 93%. 1 Οκτωβρίου, στο κλείσιμο. Το είπαμε εμεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι το τελευταίο, το, το οριστικό στοιχείο, άρα μεγάλη πρόοδο σε σχέση με πέρυσι. Επίσης, οι πληρωμές σε δόσεις από τα μέσα χρηματοδότηση για τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού θα συνεισφέρουν στο να μειωθεί ο κίνδυνο τη υποχρησιμοποιήση, τη υπεκμετάλλευση αυτών των κονδυλίων. για τις επιδόσεις, την απόδοση. Και εδώ έχουμε βελτιώσεις στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Έχουμε ένα πλήρε σύστημα πλέον υποχρεωτικών δικτών για το output και τα αποτελέσματα σε επίπεδο προγράμματος. Και όπως γνωρίζετε θα εξακολουθήσουμε να προσπαθούμε τα στοιχεία αυτά ε, για την απόδοση, για τις επιδόσεις να τα επιβάλλουμε και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ που λάβατε τα στοιχεία αυτά υπόψη και ελπίζω να τα συμπεριλάβετε και στην έκθεσή σας. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για όλα σας τα σχόλια και για τις απαντήσεις και τις δικαιολογίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένουμε όλες τις τροπολογίες. Προσωπικά θα προσπαθήσω να βελτιώσω το κείμενο με τις τροπολογίες σας. Ακόμα και αν δεν διαφωνώ και, και δεν συμφωνώ μάλλον απολύτως γιατί το 2016 υπήρξε πρόβλημα με το ορισμό και το χαρακτηρισμό. Για το 2016 μιλάμε. Αν έχει λυθεί το πρόβλημα, τόσο το καλύτερο. Επετύχαμε. Από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά εδώ πρόκειται για το 2016. Που ήταν πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ για τις προτάσεις σας και τα σχόλιά σας. Περιμένω τις τροπολογίες. Σας είπα πότε είναι η προθεσμία. 30 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι, μέρα Πέμπτη. Για να έχουμε και την ευκαιρία να ψηφίσουμε. Μάλλον Τρίτη, συγγνώμη. Στην επόμενη συνεδρίαση. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την ημερησία διάταξη για σήμερα και σας θυμίζω ότι από τις 6 και μετά ακολουθεί δεξίωση πρωτοχρονιάτικη. Και σας περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς για τη σημερινή μεγάλη μέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη. Εμείς ευχαριστούμε.